Dear colleagues, ladies and gentlemen, it's a pleasure to welcome you to this hearing on the fundamental rights implications. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Με μεγάλη χαρά σας και σας καλωσορίζω σε αυτή τη σημερινή μας συνεδρίαση για τα big data. Έχουν αυτά τα μεγάλα πακέτα δεδομένων, πάρα πολλά πλανεκτήματα για τις κυβερνήσεις και τον πολίτη. Και η Ευρωπαϊκή Στρατηγική αναγνωρίζει ω ένα μεγάλο καταδυτικό ε, παράγοντα. Δεν είναι ένα καινούριο φαινόμενο, ωστόσο η διαρκώς αναπτυσσόμενη ε, τεχνολογία με κυρίως ε, φτηνότερες και πιο προσβάσιμε λύσει, τη δυνατότητα στι εταιρείε και τι υπηρεσίε να χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο με τη δυνατότητα τα δεδομένα να συνδυάζονται ώστε να μπορούν οι ανθρώπινε συμπεριφορέ και οι πληροφορίε προσωπικέ στο μεγάλο μέρο του πληθυσμού να εντοπίζονται για σκοπού εμπορικού, επιστημονικού, υγεία και επιβολή του νόμου. Για κάποιου από αυτού του σκοπού πρέπει να πούμε ότι τα μεγάλα δεδομένα έχουν και πολλού κινδύνου. Ιδίω ό,τι αφορά την παραβίαση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, τη Ευρωπαϊκή Χάρτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Ο πολλαπλασιασμό των μεθόδων επεξεργασία των δεδομένων και τη κέντρωσή του ε, ε, από πλευρά πολλών φορέων και ανταλλαγή των δεδομένων αυτών μεταξύ του δημιουργεί τεράστια σύνορα δεδομένων που περιλαμβάνουν από τα προσωπικά για, για διάφορου είδου υπηρεσίε τα οποία τηρούνται για περιόριστο χρονικό διάστημα, ε, για πάρα πολλούς χρήστες, δημιουργώντας έτσι συσχετισμούς τα οποία μπορούν να οδηγήσουν σε αποφάσεις που μπορεί να γίνονται και με διακριτική μεταχείριση, κοινωνικές και οικονομικές επιπλοκές αποκλεισμού. Οι αρχές από τη μια και την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, έχουν εντοπίσει τι ανησυχίε του ε, σε σχέση με τα μεγάλα δεδομένα. Η έλλειψη διαφάνεια, η έλλειψη ισορροπίας και οι διακριτικές συμπεριφορές ή ε, τα διαφορετικά συμπεράσματα μπορεί να καταλήγουν στο να εκάζει κανείς διάφορες συμπεριφορές από εγκληματικέ μέχρι εκπαιδευτικέ και εμπορικές ε, για τα άτομα. Θα πρέπει λοιπόν σε όλες τις λειτουργίες των μεγάλων δεδομένων να είμαστε προσεκτικοί. Δέσμη μέτρων που εγκρίθηκε πρόσφατα ο κανονισμός με τις οδηγίες του δίνουν τη δυνατότητα ένα σύνολο κανόνων και αρχών σε σχέση με την επεξεργασία δεδομένων να διασφαλίσουν ένα υψηλό επίπεδο προστασία για του πολίτε. Ιδίω με συγκεκριμένα δικαιώματα τα οποία δεν μπορεί να αναστέλλονται. Οι κανόνε αυτέ ισχύουν για τι κυβερνήσει, για όλε τι δραστηριότητε μεγάλων δεδομένων, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτέ λαμβάνουν υπόψη και σέβονται τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ιδίω στον ιδιωτικό βίο και την προστασία των δεδομένων. Το Ευρωκοινοβούλιο στο ψήφισμά του στις 10 Μαρτίου 2016 προς μια οικονομία που την οδηγεί η συλλογή δεδομένων, τονίζει ότι οι νόμοι περί συλλογής δεδομένων πρέπει να εφαρμόζονται για όλες τις δραστηριότητες μεγάλων δεδομένων και συλλογής του την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει πλήρη συμμόρφωση. Η σημερινή ακρόαση ασχολείται με τις επιπτώσεις των μεγάλων δεδομένων στα ε, θεμελιώδη δικαιώματα εάν χρησιμοποιούνται για, ε, είτε χρησιμοποιούνται για, εμπορικές, ε, για εμπορικούς σκοπούς ή για σκοπούς επιβολής του νόμου από τις ε, αρχές. Όλοι μας οι προσκεκλημένοι θα προσφέρουν στην Επιτροπή ΛΥΜΠΕ τις απόψεις διαφορετικών φορέων από τις εταιρείε, τους καταναλωτές, τις μη κυβερνητικές οργανώσεις, τις αρχές τις διοκτικές, τις δημόσιες αρχές της ενός των πολιτών σε σχέση με το θέμα αυτό. Ελπίζουμε να έχουμε μια πολυφωνική και ευρεία κάλυψης εικόνα για αυτό το τόσο θεμελιώδες και ουσιαστικό ζήτημα. Θα ήθελα τώρα να σας παρουσιάσω τους ομιλητές, να καλέσω μάλλον τους, ε, να ευχαριστήσω τους για την αποδοχή της πρόσκλησής μας και λίγα λόγια για τη διαδικασία. Στο τέλος, κάθε μιας από, καθενός από τους δύο γύρους θα έχουμε μια φάση ρωταπαντήσεων. Επίσης να σημειώσω ότι δείτε στο διαδίκτυο αυτή η ακρόαση και ότι οι ομιλίες σας θα ηχογραφηθούν και θα μαγνητοσκοπηθούν και υπάρχει και διερμηνία. Μπορείτε να μιλήσετε ό,τι γλώσσα θέλετε. 11 γλώσσες δηλαδή. Ο πρώτος γύρος θα ξεκινήσει ευθύ αμέσω. Έχει να κάνει με την εμπορική χρήση των δεδομένων. Εδώ θα ξεκινήσουμε με τις γενικές ε, προοπτικές ε, για τα μεγάλα δεδομένα και τις σχετικές τάσεις και σε μια δεύτερη φάση θα ασχοληθούμε με τις προοπτικές των εταιριών και των καταναλωτών. Τέλος, το λόγο θα δώσουμε και στην Επιτροπή στο τέλος του δεύτερου μέρους. Γι' αυτό θα ήθελα ευθύ αμέσω να δώσω το λόγο στον εκπρόσωπο του επόπτη για την Ευρωπαϊκή Προστασία Δεδομένων, του κυρίου Ντεκούνια, ο οποίος θα μας ενημερώσει για την όλη αυτή προσπάθεια από μέρος του Ευρωπαϊκού Επόπτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, είμαι κάπω κρυολογημένο, οπότε δείξτε ενοχή για τη φωνή μου. Σα ευχαριστώ για την πρόσκληση, ευχαριστώ που με καλέσατε σήμερα. Είναι εξαιρετική πρωτοβουλία τη επιτροπή σα αυτή. Θα μπορούσατε να περάσετε στην δεύτερη διαφάνεια. Θα ήθελα μερικέ σκέψει για το τι εννοούμε με τα μεγάλα δεδομένα. Και γιατί η δική μα, ο δικός μας οφορία και όλε οι αρχέ ενδιαφέρονται τόσο πολύ για αυτό το θέμα, ω προ την τεχνολογία τα μεγάλα δεδομένα έχουν να κάνουν με τη συμπίληση δυνάμεων, τη φτηνή αποθήκευση και την διάδοση του ευρυζωνικού ίντερνετ. Η αξία για τις κυβερνήσεις και τις εταιρείες αυτών των μεγάλων συνόλων δεδομένων είναι ότι τους δίνουν τη δυνατότητα να καταλάβουν, να προβλέψουν και να σχεδιάζουν την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είναι ένα σύστημα λοιπόν ε, ιδεών και αντιλήψεων τα μεγάλα δεδομένα, πέρα από τα ίδια τα δεδομένα. Δηλαδή ότι θα μπορούσαμε με βάση αυτά να, σώσουμε οποιαδήποτε, να λυσουμε οποιοδήποτε κοινωνικο-οικονομικό πρόβλημα. Εάν όμως συλλέγονται διακρίτως και αποθηκεύονται διακρίτως, με το διαδίκτυο πώς λειτουργεί σε όλες τις χώρες, φτάνουμε να έχουμε ε, ένα τεράστιο όγκο δεδομένων. Είναι πάρα πολλοί οι φορείς πλέον που καταγράφουν ε, αόρατη τη συμπεριφορά μας. Ε, αυτό χρησιμοποιείται πολύ από τις επιχειρήσεις και αυτό είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Έχουμε τόσες διασυνδεμένες συσκευέ μεταξύ των ανθρώπων ε, στον κόσμο που αναμένεται να φτάσουμε τα 25 δισεκατομμύρια στο 2020 οι καπιταλιστές θεωρούν ότι θα φτιαχτεί το διαδίκτυο των πραγμάτων και ότι έτσι θα μπορούν να διαχειρίζονται όλη την ανθρώπινη συμπεριφορά. Όμως τα μεγάλα δεδομένα ε, έχουν δημιουργήσει προβλήματα και με την κανονική ροή πληροφοριών. Η προστασία των δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχε πάντοτε ένα διτό στόχο. Πρώτα απ' όλα, να διευκολύνουν τη ροή προσωπικών δεδομένων για να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία τη εσωτερική αγορά, αλλά προστατεύοντα ταυτόχρονα το δικαίωμα των ε, ενδιαφερομένων και τα ανθρώπινα δικαιώματά του. Πρέπει λοιπόν να διευκολύνουμε και όχι να εμποδίσουμε την χρήση των τεχνολογιών και των εφαρμογών του. Στα πλαίσια τη συζήτηση στην Επιτροπή σα, του νέου κανονισμού για την προστασία των δεδομένων και τη σχετική οδηγία, Πιστεύουμε ότι με αυτά ε, επιδιώκεται ο διεκτός αυτός στόχος. Όμως η ρομποτική, η εξέλιξη των μηχανών και η σχετική εκμάθηση επηρεάζουν πολλά από τα δικαιώματα της ανθρωπινής τη Χάρτα για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και βεβαίω κλιμακώνονται οι ανησυχίε για την προστασία. Επίση, οι πρακτικέ παρακολούθηση από τα κράτη έχουν γύρει ανησυχίε. Τώρα, οι πολίτε αρχίζουν να διρωτώνται για την υπερβολική πρόσβαση και προσπελασιμότητα από μεγάλε δεσπόζουσε στην αγορά εταιρείε. Όσοι δίνουν τα δεδομένα του, τελικά αισθάνονται ότι υπάρχει και ψηφιακή έλλειψη ισορροπία. Η μελέτη που είχε ζητήσει το Ευρωκοινοβούλιο και η Επιτροπή για τη μελέτη αυτή και για την διακριτική μεταχειρίση στι ψηφιακέ αγορέ ήταν ένα σημαντικό ορόσημο. Η έρευνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τι ΗΠΑ διαρκώ δείχνουν ότι η πλειοψηφία δεν εμπιστεύονται τι εταιρείε και έχουν αμφιβολίε για το τι συμβαίνουν με τι πληροφορίε που του αφορούν. Ιδίω με τι υπογραμμικέ υπηρεσίε. Οι πολίτε ανησυχούν διότι τα θεμελιώδη συμφέροντά του όπω αναγνωρίζονται στο πρωτογενέ δίκαιο τη Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, κλειδονίζονται. Πρώτα απ' όλα, ιδιωτικό βίο ε, παραμένει ένα αντίρρητο δικαίωμα, αλλά μπορεί να αποτελέσει και αντικείμενο διαφήμιση για γυαλιά ηλίου και για μαγιό και μπικίνι. Εδώ λοιπόν ε, Έχουμε μια σειρά από νέα φαινόμενα που παρουσιάζονται. Γι' αυτό προσπαθούμε να καταγράψουμε κάποιε αρχέ λεπτομερώ στην χάρτα, όπω τη συνένεση για την επεξεργασία των δεδομένων, την τήρηση των προσωπικών δεδομένων μετά τη συλλογή, την ελάχιστη δυνατή συλλογή, σαφήνεια για το ποιο είναι αυτό που τηρεί τα αρχεία, την σαφή περιγραφή τη επεξεργασία, τη χρήση του μόνο για συγκεκριμένου σκοπού, αυτούς για τους οποίους αρχικά συνελέχθησαν, το σεβασμό των μεγάλων ε, βασικών αυτών αρχών ακόμα και υπό μεγάλη πίεση. Ένας τρόπος να ανταποκριθούμε είναι ότι οι τεχνολογίες και οι πρακτικές αυτές απλώς είναι ασύμβατες με τις αρχέ προστασία των δεδομένων και θα πρέπει να αντισταθούμε. Μια άλλη απόκριση θα μπορούσε να είναι ότι οι αρχές μας πρέπει να μεταβληθούν για να σεβαστούμε τις αλλαγές ε, του κλίματος γύρω μας, τις αλλαγές στον καιρό μας, στην εποχή μας πρέπει να κοιτάξουμε πώ είναι όμω η πραγματικότητα των ανθρώπων αυτών που βασίζονται στα μεγάλα δεδομένα. Υπάρχει το και το θέμα τη ελευθερία τη έκφραση. Ελευθερία να επιλέξει κανεί τι περιεχόμενο θέλει να βλέπει. Ε, την έκφραση των άλλων. οι στο ιστότοποι και άλλοι τρόποι διείσδυση στον προσωπικό χώρο του καθενό, βασίζονται σε αλγορίθμους όπου προσπαθεί να παραβιαστεί ο ιδιωτικό χώρο του καθενό πολίτη. Πολλέ φορέ επιστώσει και οι ασφάλειε βασίζονται στη συλλογή ακριβώ μεγάλων δεδομένων για το υπηρεσίε προτείνοντα τους στου πολίτε. Δηλαδή, αντί να αλλάξει κάτι στο μεγάλο χέρι που ελέγχει τους πολίτες, το χέρι αυτό έχει γίνει ψηφιακό για να ελέγχονται τα τραπεζικά τους και η συμπεριφορά τους. Και είναι ενδεχόμενοι τώρα κίνδυνοι από τα μεγάλα δεδομένα, εάν δεν υπάρξουν απορροφητέ δεν θα έχουμε το κατάλληλο περιβάλλον. Θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν νόμους, κανόνες για το, εμπόριο την, για το απόρριτο και την εμπιστευτικότητα, ε, ελεγκτές και επόπτες που θα λογοδοτούν με τις ευρωπαϊκές αρχές να δίνουν το παράδειγμα. Θα πρέπει να δώσουμε την δύναμη στους πολίτες για να υπάρχει ένα σύστημα διαχείρισης που να είναι αποτελεσματικό και η μηχανική που να δίνει τη δυνατότητα για καινοτόμες λύσεις. Κατά την άποψή μας το Σεπτέμβριο φαίνεται ε, μάλλον η δική μας γνωμοδότηση διερευνά το online tracking, τη δύναμη των μονοπωλίων και το πώς ε, λειτουργούν απομονωμένα τα μεγάλα δεδομένα αλλά και το, ο οίκος εκαθάρισης ε, συμψηφισμού όπως έχει ονομαστεί των μεγάλων δεδομένων. Βλέπουμε ποιες είναι οι τιμές υποβολής για τους κοινού νόμους, ε, πρόνοια, πρόληψη κινδύνου, βιωσιμότητα και το καθεξής. Υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες σε σχέση με συνεργασίες που μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να υπάρχουν ωφέλεια τα μεγάλα δεδομένα και προστασία των πολιτών. Πάντως, βλέπουμε πώς πρέπει να συνδυάσουμε την ελευθερία της έκφρασης, ιδίω μετά την απόφαση του ΔΕΚ του 2014 και τη συζήτηση του δικαιώματος στη λύθη. Εάν δούμε και τον ιδιωτικό βίο, πώς ορίζεται στα Wikipedia ο ιδιωτικό βίος. Είναι η δυνατότητα ενό ατόμου μια ομάδα να αποκρύπτει προσωπικέ πληροφορίε και να εκφράζεται επιλεκτικά. Δεν μπορεί λοιπόν κανεί να επιβάλλει την ελευθερία τη έκφραση χωρί το δικαίωμα στη λύθη. Αυτά είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Εάν εμποδιστεί το ένα, δημιουργείται πρόβλημα στο άλλο. Λόγω χάρη μπορούν οι άνθρωποι να αποφασίσουν να χρησιμοποιούν επιγραμμικέ υπηρεσίε χωρί να το γνωρίζει κανεί και να μην παγιδεύονται. Εάν η χρήση των υπηρεσιών έχει να κάνει με συμφωνία για την χρήση δεδομένων με όρου που δεν μπορεί να διαπραγματευτεί κανεί, πριν από 10 χρόνια, ε, μάλλον είναι πολλέ οι σελίδε των όρων κάθε σύμβαση για να διαβάσει κανεί αυτέ τι λεπτομέρειε. Πρέπει να βρεθεί σωστή ισορροπία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είπε ότι υπάρχουν σοβαρέ επιπτώσει στο δίκτυο τη ενιαία αγορά. Δηλαδή, όσο πιο πολύ χρησιμοποιούν υπηρεσίε ε, οι άνθρωποι, αυτέ οι υπηρεσίε τόσο πιο πολύ γίνονται πολύτιμε και διαφημίζονται περισσότερο, ώστε τι χρησιμοποιούν ακόμη περισσότεροι. Αυτό λοιπόν έχει να κάνει με το κοινωνικό κόστος του κάποιες υπηρεσίες να μην χρησιμοποιούνται. Μπορεί να δεχτεί κανείς ότι κάποιες επιγραμμικές υπηρεσίες έχουν γίνει ουσιαστικές για την καθημερινή μας ζωή και δημιουργούν μέχρι και εξάρτηση. Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη των Αρχών για την Προστασία Δεδομένων φέτος νωρίτερα με στη χρονιά κάλεσε για την ανάγκη ενίσχυση τη συνεργασία μεταξύ των φορέων. Είναι στην εμφάνιση σα ενδιαφέρον, αλλά θα προχωρήσω στην επόμενη. Εδώ γράψαμε στους φορείς που θέλουν να συμμετέχουν σε ένα ψηφιακό οίκο ψηφισμού, εκαθαριστικό ώστε να βελτιωθεί η συνεργασία ε, μεταξύ των διοκτικών αρχών, των υπεύθυνων για την τήρηση των δεδομένων και ούτω καθεξής. Δηλαδή να υπάρχει και ένας χώρος στο διαδίκτυο που να είναι κανείς ελεύθερος από το tracking, από την καταγραφή και την εχνηλασιμότητα και να μπορεί να ασκήσει ελεύθερα το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση. Τελευταία διαφάνεια. Ήρθε η ώρα για δράση. Χρειάζονται νέα εργαλεία, αλλά πρέπει και να τα εκδιπλώσουμε μαζί καλύτερα. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Thank you very much for this... Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Και θα ακούσουμε τους εμπειρογνώμονες από τον κλάδο και να ακούσουμε τον κύριο Λουκαρίστα που εκπροσωπεί την ε, σχετική εταιρεία του Λουξεμβούργου. Θα μας παρουσιάσει τι σχετικέ εμπορικέ πρακτικέ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σα ευχαριστώ που μας ε, υποδεχτήκατε και μα καλέσατε. Είμαι ο Λουκαρίστερ ε, τη Business και Decisions Benelux. Ελπίζω να έχετε πάρει την ε, παρουσίασή μου. Να σας παρουσιάσω την εταιρεία μου. Είμαι πάροχος ε, υπηρεσιών στον τομέα του IT και αυτό που κάνουμε έχουμε 200.000 ε, consultants σε όλο τον κόσμο και παρέχουμε υπηρεσίες ε, σχετικά με δεδομένα. Συλλέγουμε δεδομένα για να ενδυναμώσουμε διαδραστικά για τις δραστικούς πληροφοριών και δεδομένων. Και ας περάσουμε στην πέμπτη διαφάνεια για να σας δείξω τι ακριβώς εννοώ. Δεδομένα λοιπόν συλλέγουμε για να μπορέσουμε να ενδυναμώσουμε τη λήψη αποφάσεων μέσω ψηφιακών καναλιών. Saying big data or small data, it's any data. Okay? So, uh, and that's... Αυτός είναι ο τομέας μας, αυτό και ειδικευόμαστε και εδώ βλέπουμε ότι έχουμε μεγάλε επενδύσει και από τον δημόσιο αλλά και τον ιδιωτικό κλάδο. Και ο σκοπό μα ασφαλώ είναι όχι μόνο η συλλογή δεδομένων, αλλά και να δώσουμε και να δυναμώσουμε τη λήψη αποφάσεων για να υπάρχει καλύτερη ε, παροχή υπηρεσιών στου καταναλωτέ και, ε, και για τις ε, πελάτε. Αυτό είναι, Αυτό είναι ο σκοπό μα. Βλέπετε κάποιου από του πελάτε μα. Δραστηριοποιούμαστε στον χρηματοοικονομικό κλάδο και εδώ φυσικά τα θέματα ιδιωτική σφαίρα είναι πάρα πολύ σημαντικά και σε δημόσιο κλάδο. Στο δημόσιο κλάδο συνεργαζόμαστε με το Υπουργείο Οικονομικών εδώ στο Βέλγιο για να αποτρέψουμε την απάτη. Εφαρμόζουμε στατιστικά μοντέλα για να προβλέψουμε, για παράδειγμα, την φοροδιαφυγή. Αυτό δίνει πολλά ωφέλη λοιπόν και συνεπάγεται πολλά ωφέλη για όλη την βαλτική κοινωνία. So, to go quick... για να δούμε την ουσία του θέματος, γιατί έκανα σύντομα την εισαγωγή μου. Βλέπουμε ότι είναι τεράστια η αύξηση στην απέτηση ε, συζήτηση για δεδομένα. Δεδομένα big data, όπως θέλετε το λέτε αλλά αυτή η αύξηση πλέον είναι πάρα πολύ σαφής. Είναι μεγάλη η μετατόπιση στη συμπεριφορά του καταναλωτή που θέλει να απελευθερώσει τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σήμερα. Επίσης, τεράστια η αύξηση για, να... για την ανάγκη αποθήκευσης των δεδομένων αυτών. Είναι μεγάλος ο ρυθμός παραγωγής δεδομένων από τις εταιρείες, όπως σας είπαμε προηγουμένως, και θέλουν όλα να φυλάσσονται να αποθηκεύονται. Αυτό έχει αλλάξει τα τελευταία δύο-τρία χρόνια, λοιπόν. Πριν από δύο-τρία χρόνια, οι επιχειρήσει προσπαθούσαν να κάνουν μια ομαδοποίηση, συγκέντρωση των δεδομένων, να διαγράψουν τι δεν χρειάζονταν. Όχι, σήμερα τα θέλουν όλα για να είναι έτοιμε για το μέλλον. Γιατί υπάρχουν πολλά παραδείγματα. Η Amazon ξεκίνησε, για παράδειγμα, να το κάνει αυτό πριν από 5-6 χρόνια, να συλλέγει τεράστιο όγκο δεδομένων αλλά πολλές ε, επιχειρήσει πλέον μιμούνται το ίδιο παράδειγμα. για να μπορούμε να κάνουμε και σύγκριση των δεδομένων αυτών. Αυτό χρειάζεται. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα δεδομένα που μπορεί να συλλέγει μια επιχειρήση, αλλά και δημόσια δεδομένα, δεδομένα τα οποία διατίθενται ελεύθερα και το web scraping, το οποίο προφανώς αποτελεί μεγάλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ιδιωτική σφαίρα και θέλουν να μπορούν να τα έχουν και να τα χειρίζονται, να παίζουν τα δεδομένα αυτά. Και επίσης υπάρχει και μεγαλύτερη ταχύτητα στην συλλογή των ε, δεδομένων. Μιλάμε για συνδεδεμένε συσκευέ, IoT κτλ. Αυτό είναι θετικό και αυτό έχουμε βάλει και θετικό πρόσημο για τις επιχειρήσεις μας, γιατί αυτό ε, συνεπάγεται πολλές καινούργιε ευκαιρίες για εμπορίο και συναλλαγές με τις επιχειρήσεις. Αλλά στην επόμενη διαφάνεια θα δείτε και κάποιους ενδεχόμενους ε, εμπόδια, κάποια ενδεχόμενα προβλήματα, γιατί υπάρχει μεγάλη παρερμηνία της νομοθεσίας. Με να οι πελάτες για το GDPR, για παράδειγμα. Για δώστε μας πληροφορίες και βοηθήστε μας Κάποιοι καταλαβαίνουν καλά τι γίνεται, κάποιοι άλλοι όχι. Υπάρχει επίσης έλλειψη πρόσφατων ικανότητων. Πολλές ε, εταιρείε, ακόμα και ιδιωτικέ, δεν έχουν και τους πόρους για να αντιμετωπίσουν αυτή τη μετατόπιση σε ό,τι αφορά, για παράδειγμα, τη συμβατότητα. Δεν υπάρχει απλά προσωπικό για να αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό για κάθε πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει δεδομένα. Επίσης υπάρχουν πολλά συστήματα επαλαιωμένα που υπάρχουν. Και εδώ και 20 χρόνια, για παράδειγμα, ε, συλλέγουν δεδομένα κάποιες επιχειρήσεις, γι' αυτό υπάρχει και δική μου εταιρεία άλλωστε. Και κάποιες εταιρείε ε, έχουν συστήματα πολύ παλιά. Επίσης, πολλοί άγνωστοι παράγοντες, όχι τόσο πολύ για την νομοθεσία, αλλά για το πώς, πώς θα πρέπει να τύχουν διαχείριση διάφορα συστήματα δεδομένων. Και εδώ δεν υπάρχει επαρκή δομή και διάρθρωση. Και βλέπουμε ότι πολλές εταιρείε σήμερα τι κάνουν. Προσπαθούν να ξεκινήσουν τη δικασία συμμόρφωσης, αλλά με έναν τρόπο κάπως άτακτο. Σαν να προσπαθούν ε, ε, βεβαιασμένα να τα πασαλείψουν όλα, χωρίς να πιστεύουν ότι μπορούν να το κάνουν με δομημένο τρόπο. Τι μας επιπλέει το μέλλον. Streaming data, IoT. Αυτό το κάνουμε ήδη. Ε, συσκευέ σε μεγάλη όγκος δεδομένων, σύνδεση, διασύνδεση με τα social media και το scraping data. Deep learning και AI σε βάθος εκμάθηση και τέχνητη νοημοσύνη. Μιλάμε για τα στατιστικά μοντέλα, τα οποία μπορούν να επεξεργαστούν τεράστιους όγκους δεδομένων, χωρίς απαραίτητα ανθρώπινη παρέμβαση. Δηλαδή, θα αρχίσουν να σκέφτονται από μόνοι του οι μηχανέ να δημιουργούν νέα αξία από τον δεδομένων. Και βλέπουμε όλο και πιο πολλέ υπηρεσίε νεφου, cloud. Αυτό είναι λίγο βαρύ για μα σε διάφορε περιστάσει, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί πάροχοι τέτοιων υπηρεσιών στο νεφο. Είναι δύσκολο να το διαχειριστούμε. Και επίση, πρόκειται για το νεφο, το cloud, και έτσι περνάνε ε, όλα αυτά τα δεδομένα από δημόσιε ε, διαδρομού και εδώ πολλά πρέπει να πάρουμε υπόψη μα. Και επίση έχουμε και νέα παραδείγματα, όπω το blockchain για τον ε, χρηματοοικονομικό τομέα. Θα γεννητομήσουν και θα διαμορφώσουν τελείω με καινούριο τρόπο το τοπίο αυτό. Τώρα κάποιε ερωτήσει, στην επόμενη διαφάνεια. Πώ θα γίνουν αυτές οι διαδικασίες πιο λειτουργικές. Privacy by design, προσωπική και ιδιωτική σφαίρα κατά το σχεδιασμό, εσείς εργάζεστε από αυτού. Είναι καλός αυτός τρόπος, ο τρόπος για να κινηθούμε για το μέλλον. Τι γίνεται και με την ε, κοινότητα GDPR, για παράδειγμα τα meetups, ε, support groups, ομάδες υποστήριξης κτλ. Εδώ νομίζω ότι ο ιδιωτικό κλάδος θα ήθελε να αναπτυχθεί περαιτέρω ο κλάδος αυτός. Να υπάρχουν πιο πολλές τέτοιες ακροάσεις, αλλά σε μορφότυπο meetup, για να μπορούμε να συζητάμε ανοιχτά τα θέματα αυτά. και τέλος πρότυπα τη βιομηχανία, ε, όπου θα υπάρχει συμμόρφωση με όλους τους ε, κανόνες. Ε. Ανησυχούμε ότι αυτή η σοκολάτα θα βγει εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου αυτό είναι δυνατόν. Επίσης μας ανησυχούν τα παράνομα έργα, τεχνικώς πώς εφικτά, εντός μιας οργάνωσης, χωρίς όμως να κινητοποιούνται στις αρχές. Και τέλος, το να κρύβεται κανείς πίσω από μικρά παραπτώματα, για παράδειγμα για να συνάδει κανείς και να συμμορφώνεται με το GPDR, θα πρέπει να ζυγίσει, ε, να συμβαδίζει με κάποιες ε, αρχές, αλλά για να κρύψει ουσιαστικά ε, μεγαλύτερα παραπτώματα. Κάποιες απαντήσεις τώρα να σας δώσουμε στη φάση των ερωταπαντήσεων θα μπορούσα να σας τα παρουσιάσω αυτά, γιατί από ό,τι βλέπω δεν έχω και πολύ χρόνο άλλο. Αν έχετε ερωτήσεις, ευχαριστώ να σας απαντήσω. Thank you very much. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίασή σας αυτή και ας περάσουμε στον επόμενο ομιλητή, τον κύριο David Martin, που εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Ένωση Καταναλωτών. Έχετε 10 λεπτά. <clears throat> Thank you very much. Ευχαριστώ. Είχα μια παρουσίαση PowerPoint, αλλά έφερα και ένα φίλο μου μαζί. Αυτή είναι η φίλη μου. Η Κέιλα. Θα την έχετε δει στις ειδήσει αυτή τη βδομάδα. Είναι μια κούκλα διασυνδεδεμένη. Θα είναι η καλύτερη φίλη της κόρης σας. Μπορεί να της μιλήσει για τα χόμπι της, για τα κατοικίδια, για το αγαπημένο της φαΐ. Είναι πολύ χρήσιμη και, πολύ και είναι και λαλίστατη. Πάντως, το Συμβούλιο μας έκανε κάποιες έρευνες για το θέμα αυτό, το, θέμα των παιχνιδιών, ιδίως των διασυνδεδεμένων και κατάφερε, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτή η κούκλα θα στέλνει τις συζητήσεις που έχει με χιλιάδες παιδάκια σε μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η εταιρεία αυτή δίνει το δικαίωμα να συγκεντρώσει αυτά τα δεδομένα για τρίτα μέρη και να τα χρησιμοποιήσει για μια σειρά από σκοπούς. Η προτεραιότητα η εταιρεία όμως είπε ότι, ότι θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την ε, πληροφορία έτσι ώστε να ε, βελτιώσουμε τις ε, πληροφορίες μας και τα δικά μας προϊόντα και επομένως θέλουμε να είναι δικά μας τα στοιχεία αυτά. Αυτή είναι Big Data Operation. Αλλά δεν είναι η Κέιλα θα έχει τη δυνατότητα να σας μιλάει, να σας λέει ποιες ταινίες ε, του Disney της αρέσει να βλέπει. Ε, βέβαια, εντάξει, έχουμε και λίγο έτσι κρυφή ε, διαφήμιση για τα παιδιά. Επίσης ε, υπάρχουν και διάφορες παραβιάσεις των αρχών της προστασίας των καταναλωτών και δεν είναι και μόνο αυτό. Ε, επίσης προωθεί η Κέιλα ε, τα στερεότυπα, τα κλισέ για τα, για τα φύλλα, δηλαδή αυτή κάνει τις δουλειές του σπιτιού, μαγειρεύει κτλ. Ε, και μάλιστα προετοιμάζουν και ένα άλλο είδος κούκλας ρομπότ που, μιλάει, που ε, είναι αγόρι και που ασχολείται μόνο με την επιστήμη και με τα πειράματα και με τα τέτοια. Ε, και επομένως καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε ε, την ε, Κέιλα η οποία, στην οποία έχουν εμπιστοσύνη τα παιδιά και η οποία, με την οποία συζητούν και δίνει στερεότυπα ε, συγκεκριμένα ε, και ε, μπορεί να δώσει και κάποιες επιπλέον πληροφορίες οι οποίες μπορεί να είναι για ομόφυλα ζευγάρια, μπορεί να είναι για διάφορα άλλα θέματα. Αυτές όμως οι λέξεις είναι απαγορευμένες. Πρέπει να πούμε ότι χιλιάδες παιδιά παίζουν με τα παιχνίδια ε, δικαιολογείται λοιπόν ε, αυτή η δυνατότητα συζήτησης ε, όχι, εγώ πιστεύω ότι δεν προωθεί καθόλου το θέμα αυτό η Κέιλα, απλώς είναι ο τρόπος, ένα παράδειγμα που δείχνει την χρήση, την δυνατότητα χρήσης των big data. Ε, ε, για την περίπτωση της ε, Κέιλα ήδη έχει αρχίσει να απασχολεί ε, τις ε, υπηρεσίες προστασίας δεδομένων ε, και στο Βέλγιο και στις κάτω χώρες. Εν πάση περιπτώσει, αν ψάξετε στο διαδίκτυο για το Toy Fail, θα σας βγάλει το παράδειγμα της Κέιλα. Τώρα όσον αφορά τα big data γενικά, εγώ δεν μπορώ να, δεν πρόκειται αυτή τη στιγμή να ασχοληθώ με όλα τα καλά στοιχεία τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ήθελα να ασχοληθώ με κάποιους προβληματισμούς, κυρίως σε σχέση με την προστασία των ιδιωτικών δεδομένων και της ιδιωτικής ζωής. Αναμφισβήτητα, οι κίνδυνοι ε, ανεβαίνουν σε τελείως διαφορετικό επίπεδο. Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος των δεδομένων και λαμβάνοντας υπόψη ότι εντός των δεδομένων το μεγαλύτερο ποσοστό ε, είναι προσωπικά δεδομένα, καταλαβαίνετε ότι υπάρχει ε, α, ε, τεράστια δυνατότητα συνδυασμού και διαχείρισης αυτών των δεδομένων και στην ουσία δίνουμε πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, τι μας αρέσει, τι τρώμε, τι δεν τρώμε, τι θέλουμε, τι δεν θέλουμε, τι ψωνίζουμε ε, και επομένως ε, με τον τρόπο ε, αυτό κάποιοι μπορούν να επηρεάσουν την συμπεριφορά των καταναλωτών. Βρισκόμαστε υπό διαρκή επιτήρηση ως καταναλωτές διαρκώς δημιουργούμε δημιουργούμε μόνοι μας το προφίλ του εαυτού μας. Κάποιοι χρησιμοποιούν αυτά τα προφίλ, ε, αντλώντας από αυτά ε, συγκεκριμένες ε, πληροφορίες, χρησιμοποιούν δηλαδή τα στοιχεία αυτά ορισμένοι, κάνοντας αλγορίθμους για να μας πούν με τι ασχολούμαστε, τι μας αρέσει, τι δεν μας αρέσει. Ξέρετε ας πούμε και είναι ένα παράδειγμα του πόσο άσχημα πάνε τα πράγματα, του ότι κάτι έγινε λάθος εάν δίνεται εάν δείτε τι γίνεται στα ε, μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά και αν δείτε ε, το Black Mirror το οποίο είναι βέβαια μια διστοπική, είναι επιστημονική φαντασία και δίνει μια διστοπική εικόνα της πραγματικότητας Εν πάση περιπτώσει, ας επανέλθουμε στην πραγματικότητα, αναμφισβήτητα το ίντερνετ των πραγμάτων και τα big data ε, λαμβάνουν υπόψη την, ε, τους ε, καταναλωτές και τους κινδύνους που παρουσιάζουν για τους καταναλωτές. Βεβαίως είναι προφανές ότι το ίντερνετ των πραγμάτων και τα big data έχουν αλλάξει τις σχέσεις ανάμεσα στις, στις υπηρεσίες και τους ε, καταναλωτές έχουν αυξήσει την έλλειψη ισορροπίας. Η ανισορροπία είναι μεγαλύτερη. Ε, οι καταναλωτές δεν ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει και ε, τι να σας πω, ε, ενδεχομένως στο μέλλον ε, δεν θα έχετε τη δυνατότητα να ασφαλίσετε το αυτοκίνητό σας παρά μόνο αν βάλετε στο αυτοκίνητο ένα μαύρο κουτί το οποίο θα δείχνει όλες τις συνήθειές σας ή ενδεχομένως για να μπορέσετε να ασφαλιστείτε όσον αφορά την υγεία σας θα πρέπει να δεχτείτε να φοράτε ένα μηχάνημα το οποίο θα ελέγχει τον τρόπο με τον οποίο κινείστε, τι τρώτε κτλ. Ε, όπως ανέφερα και προηγουμένως ε, είναι το ίντερνετ των πραγμάτων αυτό το οποίο δίνει την δυνατότητα ε, για δημιουργία ιδιαίτερα τέρος λεπτομερών προφίλ ε, καταναλωτών, τα οποία μαζί με τις αναλύσεις των big data ε, μπορούν ε, να οδηγήσουν σε προβλέψεις πολύ συγκεκριμένες. Στο μέλλον θα είμαστε ακόμα πιο πολύ στο έλεος των big data μέσω των τηλεφώνων μας, μέσω των συσκευών που χρησιμοποιούμε. Εκατομμύρια άνθρωποι ε, είναι καταναλωτές δυνάμεις σε όλο τον κόσμο και το σημαντικό λοιπόν ε, για ορισμένους ε, είναι να μπορούν να τους επηρεάσουν. Αυτό όμως επηρεάζει τη δικιά μας δυνατότητα επιλογής. Τα big data θα βοηθήσουν τις μεγάλες εταιρείες να μας υποδείξουν εν τέλει τι θέλουμε. και βεβαίως ε, ε, είτε το θέλετε είτε όχι όταν ε, κάνετε επιγραμμικά τις αγορές σας ήδη δίνετε ένα πρώτο υλικό σε αυτές τις εταιρείε, είτε το θέλετε είτε όχι κάνουν το προφίλ σας είτε το θέλετε είτε όχι. Για την ώρα είμαστε ακόμα στην αρχή και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα οδηγηθούμε. Αυτό το μαύρο κουτί στο οποίο αναφέρθηκε προηγουμένως γίνεται όλο και πιο μαύρο και όλο και πιο πυκνό και επομένως είναι πάρα πολύ δύσκολο να προστατέψουμε τις δικές μας αρχές. Ε, ε, γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να ε, δημιουργηθούν κανόνες οι οποίοι θα επιβάλλονται σωστά. Εάν παίξουμε σωστά, εάν οι κανόνες είναι σωστοί, τότε ενδεχομένως θα οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη που είναι απαραίτητη έτσι ώστε το σύστημα να λειτουργήσει καλά. Ένα στοιχείο αδιαπραγμάτευτο ως σημείο εκκίνησης είναι η προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων ε, και δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα άλλο παραπάνω. Εάν έχετε ε, παρατηρήσεις ε, μπορείτε να το κάνετε και μόλις τη σβήσετε δεν θα μπορεί να στέλνει οποιοδήποτε μήνυμα αυτή η κούκλα. Ευχαριστώ. Ωραία. Και τώρα να ακούσουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο κύριος Πολ Νίμιτς, Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση Justice, θα μα μιλήσει, Justice, θα μας μιλήσει για, την, για τις επιπτώσεις των μεγάλων στα ανθρώπινα δικαιώματα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η Επιτροπή ε, θέλει να αξιοποιήσει τα μεγάλα δεδομένα στις οικονομικές μας προσπάθειες και είναι πολύ σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ήδη ότι τα ωφέλη για τους πολίτες, είτε ως προς το εμπόριο είτε ως προς την ανάπτυξη, έχουν να κάνουν με τα μεγάλα δεδομένα. Τα οποία μεγάλα δεδομένα δεν είναι τυχαία Πρέπει να καταλάβουμε ότι κάποια μέρα όλα τα δεδομένα όλων των Ευρωπαίων θα έχουν καταγραφεί κάπου. Δεν είμαστε λοιπόν υπό την εντύπωση ότι τα προσωπικά δεδομένα είναι το μόνο θέμα που έχει να κάνει με τα μεγάλα δεδομένα, το big data, όταν μιλάμε για, το, για τα ωφέλη των πολιτών. Να μην ξεχνάμε ότι είναι πολύ σημαντικά για τις φυσικές επιστήμες, την οικονομία, τη φυσική, και είτε είναι μεγάλα δεδομένα αυτή εξ αρχή ουδέτερα που δεν είναι προσωπικά, όπω τα δεδομένα ενό μηχανήματο δεν είναι προσωπικά, είτε τα προσωπικά δεδομένα είναι ανώνυμα. Οπότε μπορούν να ε, αξιοποιηθούν πλήρω για τα δημόσια συμφέροντα <clears throat> ω μη προσωπικά δεδομένα. Εάν είναι ανώνυμα δηλαδή, δεν είναι πλέον προσωπικά. Οπότε αυτό είναι και ένας νόμος που τέθηκε σε ισχύ από τη μεταρρύθμιση της, ε, του σχετικού δικαίου. Δεύτερον, όταν μιλάμε για προσωπικά δεδομένα, τα μεγάλα δεδομένα, και αυτό είναι και η ουσία της συζήτησής μας σήμερα, ίσως όχι η καρδιά της οικονομικής συζήτησης, αλλά χρειαζόμαστε μεγάλα δεδομένα με μεγάλη εμπιστοσύνη. Μόνο έτσι μπορεί να δώσουν αποτελέσματα τα μεγάλα δεδομένα. Να το να είναι μεγάλη η εμπιστοσύνη. Αυτό το πλαίσιο θέλουμε να μας ε, επιτρέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση να δημιουργήσουμε. Κάποιες θεωρίες πηγαίνουν κατευθείαν κατά των βασικών αρχών του κανονισμού. Ορισμένοι λένε ότι η θεωρία των μεγάλων δεδομένων απαιτεί να συλλέγονται τα πάντα και μόνον εκ των υστέρων θα δούμε σε τι μπορεί να είναι χρήσιμα αυτά τα δεδομένα. Αυτό βεβαίως μπορεί να αξιοποιηθεί για να βελτιωθεί και η καμπύλη εκμάθησης. Ίσως να είναι έτσι. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι η αρχή του περιορισμού του σκοπού βάσει του άρθρου του κανονισμού, η ελαχιστοποίηση των δεδομένων, δεν μπορεί να συνάδει με αυτή την αρχή, την αρχή των μεγάλων δεδομένων. Οπότε κατά τον ίδιο τρόπο όπου δεχόμαστε ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα περιορίζουν τις δραστηριότητες σε πολλές από τις σφαίρες της οικονομικής ζωής, αλλά και όλα αυτά που εμείς κάνουμε ως άτομα περιορίζονται από άλλα κριτήρια, θα πρέπει να δεχτούμε την πραγματικότητα ότι δεν είναι όλες οι εφαρμογέ των μεγάλων δεδομένων εφικτές βάσει του κανονισμού. Θα πρέπει να έχουμε μεγάλα δεδομένα και εφαρμογέ του που συμμορφούνται πλήρως με τις βασικές αρχές. Όμως πρέπει να συμφωνούν με τον κανονισμό. Τελεία. Ο σκοπό λοιπόν εδώ είναι να υπάρχει ένα περιορισμό στο σκοπό και η ελαχιστοποίηση των δεδομένων. Είναι δυνατόν να μεγιστοποιήσουμε την δημόσια και εμπορική αξία των μεγάλων δεδομένων συμμορφούμενοι ταυτόχρονα με τον κανονισμό. Εγώ θα έλεγα ναι. Το έψαξα λιγάκι στη σχετική βιβλιογραφία και είδα ότι εταιρείε το σχολιάζουν. Οι μεγαλύτερε πολυεθνικές ουσιαστικά που συμβουλεύουν τι εταιρείε πώ να χρησιμοποιούν τα μεγάλα δεδομένα είναι η SAS λόγου χάρη λένε ότι με μια πρώτη ματιά φαίνεται ότι θα περιοριστούν οι ανάγκες ε, σε συλλογή πληροφοριών για τους πελάτες λόγω των ε, προδιαγραφών του κανονισμού και το καθεξής. Όμως, στην πραγματικότητα νομίζω ότι οι νόμοι που επιβάλλουν τη συμμόρφωση θα δώσουν μεγαλύτερε ευκαιρίε. Διότι πολλοί είναι οι οργανισμοί που επιτέλους θα πρέπει να αντιληφθούν τα δεδομένα για τους πελάτες τους στις λεπτομέρειές τους, Περισσότερο από ό,τι στο παρελθόν. Μέσω αυτής της βαθύτερης πλουσιότερης κατανόησης οι διάφοροι οργανισμοί θα καταλάβουν καλύτερα την κλίμακα των πληροφοριών, το εύρος των πληροφοριών που έχουν ήδη στη διάθεσή τους και πώς μπορούν να αξιοποιηθούν για τους σκοπούς τους. Αυτή η βαθύτερη κατανόηση θα συνοδεύεται από την ανάγκη για λογοδοσία. Την επιταγή να συμμορφούνται κανείς και με αυτή την ανάγκη. Οπότε, Θα πρέπει να υπάρχει σαφή διαχείριση και διακυβέρνηση. Οργανισμοί συμμόρφωση θα καταλάβουν ότι χρειάζονται το απαραίτητο επίπεδο εκτελεστική υποστήριξη για να χειριστούν τα δεδομένα των ε, πελατών του και νομίζω ότι αυτή ήταν και η άποψη τη SAS ότι αυτό θα είναι το μόνο θετικό. Μόνο θετικό, αλλά μπορεί να είναι για του αναλυτέ δεδομένων. Να προσθέσω εδώ ότι πολύ συχνά το ίδιο θα συμβαίνει και όταν αφορά την επιβολή του νόμου. Μαθαίνουμε τώρα ότι πολλές αστυνομικές δυνάμεις πνίγονται στα δεδομένα. Οι βασικές αρχές που τίθενται στους νόμους προστασίας των δεδομένων από το 1995, ότι τα δεδομένα πρέπει να είναι ακριβή, πρέπει να είναι επίκαιρα, πρέπει να είναι σκόπιμα. Όλα αυτά είναι αρχές που χρησιμοποιούνται για τις αρχές στα συλλογή δεδομένων τους. Οπότε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Είμαστε πλήρω ε, συνειδητοποιημένοι για τη συλλογή δεδομένων και προηγουμένω, όταν επεξεργαζόμασταν την οδηγία και τον κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην εργασία της, των διεκτικών αρχών, των αρχών επιβολή του νόμου, νομίζουμε ότι μπορούμε να έχουμε τεράστια ωφέλη και για τη δημόσια ευημερία, αλλά και για σκοπούς άλλους εμπορικούς και πολλούς ακόμη. Να αναφέρω κάποιου τιμής όπου τα μεγάλα δεδομένα, ακόμη και αν χρησιμοποιούνται σε συμμόρφωση με τους βασικούς νόμους, μπορεί να έρχονται σε αντίθεση με, την, με άλλα θεμελίδια δικαιώματα. Το ΔΕΚ ανέφερε στη σχετική του απόφαση για την ευθερία της έκφρασης. Εγώ να αναφέρω και την ελευθερία του συναφρίζεστε τη κυκλοφορία των ελεύθερων και ουδέτερων ανεξάρτητων εκλογών. Διαβάζουμε ότι στην τελευταία εκλογή του Πρόεδρου Ομπάμα ο νικητή νίκησε λόγω τη υψηλή ποιότητα των κυκλομετρικών προφίλ των ψηφοφόρων του. Ποιο είναι ο αντίκτυπο των μεγάλων δεδομένων στη δημοκρατία, διακριτική μεταχείριση βεβαίω κατά πρώτον. Και μετά ε, νόμοι εργατικού δικαίου. Σε όλους αυτούς τους τομείς θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, να καιροφυλακτούμε, διότι όπως έλεγα τα μεγάλα δεδομένα θέλουν και την μεγάλη εμπιστοσύνη των πολιτών, των εταιριών, των κρατών, των βουλευτών. Η αρχή αυτή δεν έχει να κάνει μόνο με την προστασία των προσωπικών δεδομένων, αλλά και με την πίστη ότι τα μεγάλα δεδομένα δεν θα πιέσουν αρνητικά τα υπόλοιπα δικαιώματα. Από την σκοπιά των θεμελιών δικαιωμάτων, νομίζω ότι τα περιέγραψα όλα αυτά και θα ήθελα να ολοκληρώσω λέγοντα ότι το να διασφαλίσουμε αυτέ τι βασικέ ελευθερίε και τι πραγματικά ε, δημοκρατικέ και ελεύθερε εκλογέ, η ελευθερία του εκφράζεστε, του συναθρίζεστε, τη κυκλοφορία, κυκλοφορίας, το να γνωρίζει κανεί τι συμβαίνει με τα δεδομένα του όταν συλλέγονται παντού τον κόσμο, με αναλυτέ δεδομένων παντού γύρω μα, όλα αυτά δεν είναι μικρές τεχνικές προκλήσεις, είναι ζητήματα καθοριστικά που θα διαμορφώσουν την έννοια της ελευθερίας και των θεμελιωδών δικαιωμάτων στην ψηφιακή εποχή. Ευχαριστώ. Thank you. Σας ευχαριστούμε κύριε Νίμιτς. Και μετά τις ε, τέσσερις αυτές παρουσιάσεις για το θέμα αυτό της εμπορικής χρήσης και αξιοποίησης των ε, Big Data, των μεγάλων πακέτων δεδομένων, θα ήθελα να ανοίξω το βήμα και να ακούσουμε τους ε, ομιλητές μας, να ακούσουμε τους βουλευτές μας με ερωτήσεις. Ε, να ξεκινήσουμε με την εισηγητρία, την κυρία Γκόμες. Και μετά να ακούσουμε και τους υπόλοιπους. Θα σας ζητήσω να περιοριστείτε σε δύο λεπτά, προκειμένου να έχουν και χρόνο οι ομιλητές μας να απαντήσουν. Η κυρία Γκόμες, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσες και προκλητικέ σχεδόν οι παρουσιάσει σα και οι προειδοποίησει που μα απευθύνετε. Για μα είναι σαφέ ότι το GDPR αποτελεί ένα βασικό πυλώνα που θα πρέπει να διατηρήσουμε και αποτελεί και ένα βασικό στοιχείο εμπιστοσύνη, ε, Την εμπιστοσύνη που μόλις ανέφερε ο κύριος Νέμιτς. Να ρωτήσω λοιπόν τον κύριο Ρίστερ το εξή. Ανέφερε ένα κίνδυνο. Οι εταιρείε όπω η δική του να εκλείψουν από την Ευρώπη ο λόγω των περιορισμών που επιβάλλονται από το GDPR. Όταν πέρασε όμως το GDPR αυτό ο κανονισμό για την προστασία γενικών δεδομένων, ε, ήταν σαφέ, ε, για παράδειγμα, στη ΣΥΠΑ και αλλού, ότι ήταν απαραίτητο αυτό ο κανονισμός, ιδάλλοντας δεν θα υπήρχε βιώσιμη, ε, βιώσιμος κλάδος στον τομέα αυτό. Πείτε μου λοιπόν συμφωνείτε και ήθελα να ακούσουμε και τον κύριο Ντουκούνια και τον κύριο Μάρτιν. Τι έχετε να μα πείτε για τον ενδεχόμενο κίνδυνο διακριτική μεταχείριση, Πώ μπορούμε να εντοπίσουμε τους παράγοντες κινδύνου. ακόμα και αν τα δεδομένα είναι διαμορφωμένα με ανώνυμο τρόπο. Πάντα μπορούν να επανασυνδεθούν στο άτομο. Μπορεί να αντιστραφεί δηλαδή αυτή η διαδικασία ανωνυμοποίησης. Πείτε μας επίσης πώς ένα άτομο πώς μπορεί ένα άτομο να ελέγχει τα δεδομένα του. πώς μπορεί να λαμβάνει αυτόνομες αποφάσεις, ανεξάρτητες αποφάσεις και να ελέγχει κάποια από τα δεδομένα αυτά. Δεδομένη και τη περιπλοκότητα του αντικειμένου και του γεγονότο ότι είναι πολύ αναλφάβητη ψηφιακά οι πολίτε σε πολλέ περιπτώσει. Αυτά επί του παρόντος. Ευχαριστώ, λέει ο πρόεδρο. Η κυρία Σίπελ. Σα ευχαριστώ. Και θα ήθελα καταρχά να συμφωνήσω με τον Πάουλ Νέμιτ. Ε, τα μεγάλα δεδομένα θα μπορούσαν να είναι μεγάλε μηχανέ δεδομένων, το οποίο θα μπορούσε να βοηθήσει, για παράδειγμα, αν έχουμε στι ε, δρόμου ε, αισθητήρε, οι οποίες ε, μπορεί να μας ειδοποιούν όλες αυτές τις συσκευές πώς να αποφεύγουμε ατυχήματα, μπλοκαρίσματα κτλ. Από την άλλη υπάρχει και ο δυτικός κλάδος ε, για τα μεγάλα δεδομένα. Όταν το στο κινητό μου, για παράδειγμα, το αυτοκίνητό μου συλλέγει δεδομένα για το πώς επιταχύνω, πώς οδηγώ, πώς φρενάρω. Αυτά είναι δεδομένα τεχνικά. Αλλά όταν το πάω στο εργαστήριο, όταν το πάω στο γκαράζ το αυτοκίνητό μου, μπορεί να παρακολουθεί τελικά το γκαράζ πώς οδηγεί η κυρία Σίπελε. Και ξέρουμε ότι αυτό μπορεί να έχει διάφορε συνέπειε. Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Μάρτιν που έφερε την κούκλα αυτή μαζί, γιατί μα έδειξε με σαφή τρόπο ότι το θέμα δεν είναι μόνο η συλλογή των δεδομένων και η ερμηνεία, η χρήση με οποιοδήποτε τρόπο των δεδομένων αυτών, αλλά ότι αυτή η κούκλα δίνεται σε ένα παιδί και ο παραγωγός δεν έχει στοιχεία για το παιδί αυτό πράγματι και παρόλα αυτά συλλέγονται και χειραγωγούνται πολλά στοιχεία. Και φυσικά αυτό δεν θα είναι πάντα ε, και δεν είναι υπέρ του συμφέροντος του παιδιού. Όχι. Υπέρ εμπορικών σκοπών θα γίνεται αυτή η χειραγώγηση. Άρα η καπιταλιστική αυτή αξιοποίηση διάφορων τομέων της ζωής σε διάφορα επίπεδα είναι ανησυχητική και θυμάμαι ότι ο αρμόδιος επιτροπός είχε πει πρόσφατα ότι οι ηλικιωμένοι, οι οποίοι είναι μόνοι τους στο σπίτι, μπορούν να συνομιλούν με ένα ρομπότ. Για μένα αυτό προσωπικά αποτελεί καταστροφή. Εγώ, άμα γυράσω, όχι μόνο θα ήθελα να έχω έναν άνθρωπο δίπλα μου, αλλά μπορεί να μου προγραμματίσουν ένα ρομπότ να μην τσακώνεται ποτέ μαζί μου. Ξέρετε, θα τρελαθώ άμα δεν μου μιλάει ποτέ κανείς. Άρα λοιπόν θα πρέπει να σκεφτούμε πού χρειάζεται και πού δεν χρειάζεται και πού πρέπει να ρυθμιστεί η συλλογή δεδομένων. Κάτι τελευταίο να πω. Αν μπορεί ένα προϊόν να διαπιστώσει ποιος μένει που μόνος του για πόσο πλένεται, πόσο συχνά πλένεται και πόσο συχνά κάνει ντους ή κατά πόσον ε, μπορεί να ρυθμίζει ο πάροχος ε, ενέργειας, ε, πόση ενέργεια, σε ποια φάση της ημέρας, όλα αυτά τα όρια είναι πολύ λεπτά και ρευστά. Αλλά πέρα από όλα αυτά, πίσω από όλα αυτά, είναι η ιδιωτική σφαίρα του ατόμου και αυτή διακυβεύεται και αυτό κανείς δεν μπορεί να το αμφισβητήσει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Επόμενος μιλητής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και είμαι βέβαιος ότι θα φτιάξουμε και τη κυρία Ζήπελ ένα ρομπότ το οποίο να διαφωνεί μαζί τη και να τη βγάζει γλώσσα. Θα τη το δώσουμε τα επόμενα Χριστούγεννα, δεν υπάρχει θέμα. Για δώρο. Μία από τι ερωτήσει που ήθελα να θέσω για όλα τα θέματα με τα δεδομένα αυτά. Ναι, πρέπει να δώσουμε στους καταναλωτές ε, την τελική απόφαση για να συνενέσουν ή να μην συνενέσουν. Αλλά στην τελική ανάλυση μπορεί να μην ενδιαφέρονται οι Καταναλωτέ. Ε, αν, για παράδειγμα, έχει κανεί να αναβαθμίσει το λογισμικό του, ε, αναβαθμίσει το iPhone πριν από λίγο καιρό. Ε, εννοείται ότι επιλέγω το πεδίο στο τέλο, σύμφωνα με τους ε, όρου ε, και τι συνθήκε που προβλέπει η εταιρεία. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά ζητήματα για το μέλλον, θεωρώ. Όχι μόνο του δίνουμε τη δυνατότητα να, να δίνουμε τη δυνατότητα να συνενούν ή όχι, αλλά και πώς μπορούμε αυτές οι πληροφορίες να είναι και προσβάσιμες προκειμένου να καταλαβαίνει ο κόσμος τι είναι αυτό που υπογράφει και εγκρίνει. Και νομίζω ότι αυτό θα γίνει όλο και πιο σημαντικό. Να δοθούν ε, έξυπνες λύσεις για να υπάρχει πρόσβαση σωστή στα δεδομένα αυτά. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτά που είπε ο κύριος Ρίστερ, πείτε μας λίγο πώς τα χρησιμοποιείτε τα δεδομένα και τι δεδομένα χρησιμοποιείτε για να καταπολεμήσετε τη φοροδιαφυγή, για να βοηθήσετε τις αρχές στην καταπολέμηση της απάτης. Τι δεδομένα συλλέγεται. Ποιο είναι το περιβάλλον προστασίας δεδομένων όπου χρησιμοποιείται τα στοιχεία αυτά. Και τώρα για να επανέλθουμε στο παράδειγμα της κούκλας. Νομίζω ότι ο κύριος Μάρτιν είπε ότι οι, οι όροι παραβιάζουν διάφορου νόμου για την προστασία του καταναλωτή. Πώ γίνεται λοιπόν να περνάνε αυτοί οι όροι. Και μία ερώτηση προ όλου του ομιλητέ. Τι αισθάνεστε για την... Πώς, τι πιστεύετε μπορούν οι αρχές επιβολής του νόμου να επιβάλλουν πραγματικά την νομοθεσία αυτή και το πακέτο προστασίας το οποίο εγκρίναμε, πώς πιστεύετε ότι θα συμπεριφερθεί σε σχέση και με τις μελλοντικέ εξελίξεις. Είμαστε καλά για κάποια χρόνια τώρα. Και ο τρόπος που καταρτίζουμε την νομοθεσία μας σε ευρωπαϊκό επίπεδο πιστεύετε ότι είναι κατάλληλος για να παρακολουθήσει τις εξελίξεις ε, και τις αλλαγές στον ψηφιακό κόσμο. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Και τελευταίος ομιλητής, η κυρία Λεωστίνη. Thank Σας ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους τους ομιλητές γιατί ήταν ε, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ήταν μεγάλη παρουσίαση και μάλιστα με διαφορετικές απόψεις. Εγώ πάλι έχω και άλλη διαφορετική άποψη. Εμείς 40 ε, χρόνια πριν ε, που ήμουν φοιτήτρια προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τον κόσμο με διαφορετικό τρόπο και καταλαβαίναμε αυτά που ε, μας περιτριγύριζαν με τη χρήση των ματιών μας, των αυτιών μας και του στόματός μας και τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Βέβαια αυτό που είναι νέο είναι η ταχύτητα, είναι επίσης το μεγάλο ποσοστό δεδομένων που μπορεί να χειριστεί ε, μία μηχανή και να τα αποθηκεύσει γιατί βεβαίως ε, ε, ε, οι εγκέφαλοι μας μπορεί να έρχονται σε επαφή ο ένας με τον άλλον, αλλά δεν μπορούν να αποθηκεύσουν τέτοια στοιχεία με τα big data. Στην ουσία εμείς αποκαλύπτουμε κάποια πράγματα τα οποία ήταν κρυμμένα στην, στον πολιτισμό μας, άρα θα πρέπει στην κουλτούρα μας, άρα θα πρέπει να προσαρμόσουμε την κουλτούρα ε, κοιτάξτε, ε, ε, δημιουργούμε λέξεις. αυτό το CDRP είναι μία λέξη, είναι μία γραμματική κατασκευή, αλλά η γραμματική κατασκευή δεν θα βοηθήσει από μόνη της. Άρα εδώ είναι το ερώτημα. Πώς θα υλοποιήσουμε πώς θα επανακωδικοποιήσουμε την πραγματικότητα έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στην νέα κουλτούρα. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να δώσουμε και περιεχόμενο. Εσείς ε, ο κάθε ένας από σας, ε, έδωσε μία διαφορετική έννοια εγώ δεν μπορώ να συμφωνήσω πλήρως ούτε με τον ένα, ούτε με τον άλλον, ούτε με τον τρίτο, αλλά παρόλα αυτά κάθε φορά ε, ε, ε, παίρνω κάποια στοιχεία από τον καθένα σας. Και όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά έτσι ώστε κυρίως να καταλάβουμε με ποιο τρόπο θα πρέπει να νομοθετήσουμε επιπίου θέματος θα πρέπει να νομοθετήσουμε. Ε, ε, εγώ δεν λέω ότι θα πρέπει να επανεφεύρουμε τον τροχό. Ε, ή ας πούμε λέω ότι ε, θα πρέπει αν έχουμε ένα κρίσταλο να το κρατήσουμε σε καλή ποιότητα και διαφανές γιατί εάν του βάλουμε στοιχεία τα οποία δεν θα είναι σωστά τότε δεν θα κρατήσει τη διαφάνειά του το κρίσταλο. Τώρα, τι να σας πω τώρα, αν αυτή, αυτή η κούκλα που μας δείξατε ε, δεν είναι σωστή και ότι μπορεί να δείξει ότι τα αγόρια κάνουν χι δουλειές και τα κορίτσια κάνουν ψι δουλειές, Εγώ δεν συμφωνώ και απολύτω με αυτό, γιατί όταν είσαι δύο χρονών παιδάκι, ε, ίσω χαίρεσαι πολύ που ανακαλύπτεις αν είσαι αγόρι ή αν είσαι κορίτσι. Το ζήτημα είναι ε, να υπάρχουν οι κανόνες προστασίας των καταναλωτών. Στην ουσία δηλαδή, στην, στην ουσία ήδη, ήδη τώρα είναι παράνομο τις αρχές που διέπουν το σπίτι σου να τις δώσεις, να τις παραχωρήσεις ε, σε μια εταιρεία. Τα νέα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε. Ε, τα νέα πράγματα επί των οποίων δεν έχουμε νομοθετήσει. Δεν έχουμε δηλαδή σαφώς διατυπωμένες αρχές και νόμους για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει και κάτι άλλο που σχετίζεται με τα big data. Ε, το όριο ανάμεσα σε προσωπικά και μη προσωπικά ε, μεγάλα δεδομένα δεν είναι σαφές. Ε, ας πούμε υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία στην αρχή ήταν συλλογικά δεδομένα ε, και, και δεν ήταν ε, προσωπικά, ενώ σιγά σιγά άλλαξαν στο GDPR νομίζω ότι αναφέρονται αυτά, αλλά άλλο η θεωρία και άλλο η πράξη. Στην πράξη τα πράγματα μπορεί να είναι πολύ διαφορετικά. Πρέπει να καταλάβουμε σαφώς ποιες είναι ε, ε, ποια είναι τα περιβάλλοντα επί των οποίων δεν έχουμε δικαιοδοσία ποια είναι τα θέματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε καταλάβει καν ότι είναι προβληματικά. Ε, εδώ χρειάζεται και παιδαγωγία, χρειάζεται εκπαίδευση. Εδώ φαντάζομαι ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ε, οι οποίοι χρησιμοποιούν συνεχώς τα στατιστικά ε, στοιχεία στην καθημερινή τους ζωή. Ε, και εγώ το κάνω. Αλλά τώρα το να πεις αυτούς τους ανθρώπους ότι χρειάζονται διαφανείς αλγόριθμοι είναι κάτι που τους ξεπερνάει. I now give the floor back to the speakers um, and. Uh, πάρα πολύ ωραία. Τώρα, α, Άννα, Άννα ε, θέλω μερικές ερωτήσεις ακόμα στον κύριο ε, Βίτσα σε σχέση με αυτά που είπε ότι δηλαδή μπορεί να υπάρχουν κρυφά σχέδια και ότι ενδεχομένως θα υπάρχει κάποια, ε, κάποιος πειρασμός να κρυφτεί κανείς πίσω από μικρές ε, ε, κυρώσεις έτσι ώστε να κάνει μεγάλες παραβιάσεις. Ξέρετε κάποιες τέτοιες περιπτώσεις, ε, ε γνωρίζετε περιπτώσεις όπου χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένε τεχνικές έτσι ώστε να οδηγήσουν ας πούμε σε διακριτική μεταχείριση ε, ή σε ε, ε, τραπεζικές λειτουργίες. Ε, ε, ρωτώ δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένες περιπτώσεις από τις οποίες μπορούμε να μάθουμε κάποια πράγματα, να ξέρουμε πώς να προφυλαχτούμε, να ξέρουμε πώς να προσαρμοστούμε να ξέρουμε πώς να νομοθετήσουμε έτσι ώστε ο αντίκτυπος να είναι όσο γίνεται λιγότερο σοβαρός. Ευχαριστώ πολύ. Θα επανέλθω λοιπόν στους ομιλητές. Ο καθένας μπορεί να απαντήσει μέχρι τέσσερα λεπτά και αν είναι δυνατόν να απαντήσετε συγκεκριμένε ερωτήσει που απευθύνθηκαν. Ευχαριστώ πολύ. Ε, δεν ήμουν στόχος των ε, περισσότερων ερωτήσεων και δεν τις άκουσα κιόλας όλες, αλλά θα απαντήσω σε μερικές. Κυρία Γκόμες, ρωτήσατε ε, ε, κάτι για το θέμα της διακριτικής ε, μεταχείρισης των διαχωρισμών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο άρθρο 15H αναφέρεται ρητά ότι το άτομο έχει το δικαίωμα ε, να ε, κατανοήσει την λογική της, ε, του χειρισμού και της επεξεργασίας των δεδομένων και ότι τα μεμονωμένα άτομα έχουν την δυνατότητα να μελετήσουν τους αλγορίθμους και ενδεχομένως ορισμένες περιπτώσεις να αντιταχθούν σε αυτούς. Βεβαίως το θέμα δεν μας ενδιαφέρει, που μας ενδιαφέρει δεν είναι μονάχα το νομοθετικό, μας ενδιαφέρει ο σχεδιασμός των επιγραμμικών ε, υπηρεσιών ε, και ο τρόπος με τον οποίο αυτοί προωθούνται. Και πολύ ωραία τα απεικόνισε ε, ο Ντάβιντ με την κούκλα του. Ερωτήσεις για το GDPR να σας πω ότι δίνει όντως πολλές ε, υπευθυνότητες, ε, ε, αρμοδιότητες συγγνώμη, στις αρχές εποπτείας των δεδομένων στην ομάδα εργασίας του άρθρου 29 προσπαθούμε να βρούμε μια καλύτερη ανταπόκριση ε, των ε, εποπτικών αρχών. Προσπαθούμε να καταλάβουμε, να δώσουμε στους ε, επιτηρητές των δεδομένων να κατανοήσουν καλύτερα τα πράγματα. Πρέπει να είναι προετοιμασμένοι και να έχουν τους απαραίτητους πόρους έτσι ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν. συζητούσαμε έναν συνάδελφο της, από την DPA, και μου έλεγε, αναφέρθηκε στους νέους κανόνες της GDPR που δεν τους ε, γνωρίζουμε ακόμα καλά ε, και ε, Ε, ο Τζοβάνι Μπουτσαρέλη έλεγε επίση ε, ότι το θέμα δεν είναι να έχουμε νόμους αλλά να λειτουργούν καλά. Νομίζω ότι το 2010 ξεκίνησε η διαδικασία για την οδηγία προστασίας των δεδομένων ε, και θα αρχίσει να εφαρμόζεται πλήρως το 2018. Καταλαβαίνετε 8 χρόνια έτσι ώστε να προετοιμαστεί αυτός ο νόμος. Τέλος. Πολύ ενδιαφέρον αυτό που είπε η τελευταία ομιλήτρια. Είχαμε μια συνάντηση με τον ε, νέο ε, διευθυντή της Υπηρεσίας Θεμελιωδών Δικαιωμάτων πρόσφατα ε, και μιλήσαμε σχετικά με την νέα του θέση και το κύριο στοιχείο που ανέφερε είναι ότι θα πρέπει να, σταματάμε, να σταματήσουμε να μιλάμε για δικαιώματα και για νόμους αλλά να μιλάμε πλέον για την, τον αντίκτυπο συμπεριφορών, των συμπεριφορών ας πούμε των μεγάλων εταιριών. Αυτό θα πρέπει να το σκεφτούμε και όσον αφορά την ε, προστασία δεδομένων, γιατί μπορεί να χρησιμοποιούμε πολλούς ειδικού όρους, αλλά το θέμα παραμένει απλό όσον αφορά δηλαδή τον αντίκτυπό του, τι συμβαίνει στην αγορά και κατά πόσον ε, τα όσα συμβαίνουν στην αγορά έχουν επίπτωση στην καθημερινή ζωή όλων μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ να απαντήσω σε κάποιες από τις ερωτήσεις. Ε, δεν ήθελα να είμαι ο βασικός αντίπαλος του Bring All, Use All. Δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου. Κοιτάμε στην παρουσίαση πού πάνε πράγματα, ποιε είναι οι τάσεις. Το privacy by design είναι διαφορετικό από αυτό το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε με τους πελάτες μας. Η πρώτη ερώτηση τη κυρία Γκόμε. για τις ε, εταιρείε ε, που βγαίνουν εκτό Ευρώπη. Αυτό ισχύει για τι δικέ μα εταιρείε, γιατί είμαστε πάροχο υπηρεσιών. Μπορεί να υπάρχουν και παγκόσμιοι όμιλοι οι οποίοι έχουν σε όλες τις χώρες ε, εταιρείε. Για παράδειγμα, πληρώνει κανείς ε, αγοράζει κανείς κάτι στην εταιρεία αυτή στο Μαρόκο, αλλά η πιστοτική εταιρεία, για παράδειγμα, είναι από την Ισπανία. Τι ζείτε εδώ πέρα. Είναι λεπτή η γραμμή του που βρίσκονται τα δεδομένα. Στην περίπτωση αυτή χρειάζονται και χρησιμοποιούνται ενδεχομένω δημόσια ειδικά ανέφη για την αποθήκευση των δεδομένων. Και αν αρχίσουμε να εμποδίζουμε τι εταιρείε αυτέ λέγοντα ότι τα δεδομένα πιστοτικών καρτών δεν μπορούν να τηρούνται εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα σε ό,τι αφορά τα οποία, για παράδειγμα, δεν μπορούν να τηρούνται τα δεδομένα αυτά στην Ευρώπη. Αλλά υπάρχουν θηγατρικέ στην ε, Ευρώπη και τι θα γίνει, ενδεχομένω να χρησιμοποιήσουν το ιδιωτικά του νεφι για να τα φυλάσσουν τα στοιχεία αυτά και να φύγουν οι εταιρείε αυτέ από την Ευρώπη. Αυτά σε ό,τι αφορά το νέφος υπάρχουν πάρα πολλέ τεχνικέ τεχνικές Σε ό,τι αφορά περιπτώσεις απάτης και διακριτικής μεταχείρισης. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ PIA παντού σε ό,τι αφορά τα δεδομένα. Δηλαδή προσωπικά στοιχεία τα οποία μπορούν να εντοπιστούν, να ταυτοποιηθούν σε πολλές περιπτώσεις. ίσως να μην υπάρχονται όμως στο GDPR, στο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων. Και αν γίνει σύνδεση με νέα παραδείγματα όπως το big data, το streaming data, αυτός ο κλάδος είναι όλο και πιο μεγάλος, γίνεται όλο και πιο μεγάλος. Γι' αυτό λοιπόν το θέμα των κληροδοτούμενων συστημάτων, των παροχημένων συστημάτων, τα οποία εξακολουθούν να υφίστανται στις εταιρείε σε κάποιες περιπτώσεις. Μία ερώτηση τώρα έγινε και για το πώς ε, μπορεί, για παράδειγμα, εντοπιστεί η ενδεχόμενη απάτη. Δεν είναι ο μοναδικό μα πελάτη στο Υπουργείο Οικονομικών. Υπάρχουν διάφορα δεδομένα στι αγορέ και έχουμε πολλού ε, επιστήμονε, στατιστικολόγου, ε, μαθηματικού ε, που αναπτύσσουν μηχανισμού στατιστική και του συνδέουν με τα δεδομένα των πελατών. Τα συνδέουν ενδεχομένω και με τα social media και έτσι λειτουργούν οι μηχανισμοί αυτές. Και επίσης τώρα πολλές εταιρείες σκέφτονται να μπουν και στα κοινωνικά δεδομένα, όπου ο κόσμος ε, κατά δημοσιεύει κάποια δεδομένα, προκειμένου να εμπλουτίσουν τα μοντέλα για την ανάλυση ενδεχόμενης απάτης και κινδύνου, για να μπορούμε να τα δυναμώσουμε όλα αυτά με την εμπειρογνωμοσύνη μας. Για τη τα μεταχείριση, όχι, όχι. Εδώ όχι. Ξέρω ότι υπάρχουν ε, κάποιες περιπτώσεις online ε, βάσει τεχνητής νοημοσύνης και βάσει διαφόρων μελετών μηχανισμών που προτείνουν προϊόντα από χαμηλότερες ή από υψηλότερες τιμές ανάλογα με την ανάλυση που κάνουν για τα άτομα. Αυτό έχει να κάνει με τα μοντέλα τα οποία δημιουργούνται και κατά πόσο να ακολουθούν την ανθρώπινη λογική ή όχι. Ευχαριστώ πολύ, David Martin. Σας ευχαριστώ πολύ και καταρχάς θα ήθελα να διευκρινίσω ότι το μήνυμά μου δεν είναι ότι τα πράγματα βρίσκονται σε καταστροφική φάση και ότι είμαστε καταδικασμένοι. Όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξή, ότι αν ξεχάσουμε τι θεμελιώδει μα αξίε και αφήσουμε τι οικονομικέ πτυχέ και τα εμπορικά συμφέροντα να επικρατήσουν, ενδεχομένω να καταλήξουμε σε μια πολύ δύσκολη θέση. Αυτό προσπάθησα να πω. Ακούσαμε κάποιες ερωτήσει ε, σε ό,τι αφορά το θέμα της διακριτικής μεταχείρισης. Ε, μα το ανέφερε ο συνάδελφο. Αλλά, για παράδειγμα, ακούσαμε ότι ανάλογα με τον υπολογιστή που χρησιμοποιεί κανεί η τιμή που βλέπει για ένα προϊόν κανείς σε, μια ιστοσελίδα είναι διαφορετική τα big data που θα μας επιτρέψουν ωστόσο να φτάσουμε στο σημείο του να ξέρουμε τι κοστίζει κάτι για μένα τώρα. Γιατί θα λάμβανε υπόψη στην περίπτωση αυτή του μοντέλου αυτό διάφορες παραμέτρους. Πού πήγε κανείς ε, και μπορεί να πάει κανείς ε, σε ένα μαγαζί και να μην έχει καν τιμή το προϊόν. Απλά να αναφέρεται στο τηλέφωνο του, του καθενό. Πόσο κάνει για το συγκεκριμένο άτομο τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή το προϊόν. Και σκεφτείτε τι γίνεται όταν προσπαθείτε να αγοράσετε ένα εισιτήριο αεροπορικό και αναρωτιέται κανεί μήπω πρέπει να έχει βρει τα κούκκι του και γιατί η τιμή διαφέρει τόσο πολύ από την τελευταία φορά που την κοίταξε. Ένα άλλο θέμα είναι πώς μπορούν να λαμβάνονται ανεξάρτητες αποφάσεις όταν κανείς δεν έχει εξουσία. Η μοναδική απάντηση που υπάρχει πολύ φοβάμαι είναι ότι δεν μπορεί κανείς να λαμβάνει ανεξάρτητες αποφάσεις. Δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ή το παίρνει το αφήνει. Δεν είμαστε ενήμεροι. Επαναλαμβάνω το πώς δουλεύει το κάθε προϊόν. Και γι' αυτό σας λέω ότι αυτό αλλάζει την θεμελιώδη σχέση μεταξύ υπηρεσιών, μάλλον παρόχων και πελατών. Ξέρω για παράδειγμα ότι ο φούρνο ε, μου ψήνει ψωμί, το ράζω, βγάζει χρήματα. Είναι πολύ πιο δύσκολο να καταλάβω τι κάνει η επιχείρηση του διπλανού μου. Ένα άλλο θέμα που είναι ενδιαφέρον για του καταναλωτέ. Δεν ε, σα τα κάνουν ε, για να για να τα καταλάβετε. Αν σα είχαν δύο παραγράφου αντί για εννιά σελίδε, ε, θα τα διαβάζετε ενδεχομένω. Και αν ήταν και κατανοητά, θα το διαβάζετε ακόμα πιο πιθανό, γιατί να σα πω και κάτι άλλο. Και να δώσετε το χρόνο που χρειάζεται για να διαβάσετε τι 9 σελίδε, δεν θα καταλάβετε και πάλι. Και να καταλάβετε επίση δεν έχετε επιλογή. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σα, άρα θα αποταθείτε του όρου τη Apple. Το σύστημα λοιπόν λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί να επιτρέψει πραγματική επιλογή. Και αυτά πρέπει να αλλάξουν, θεωρούμε. Και να αναφέρω και κάτι άλλο. κοιτώντα το ευρωμαρόμετρο και όλε αυτέ τι μελέτε, αυτό δείχνει ότι ο κόσμο ενδιαφέρεται για τα πράγματα αυτά. Αν μιλήσετε στον κόσμο για την κούκλα, άμα βγείτε στον έξω κόσμο, θα πείτε ότι υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον, αλλά πολλά ακόμα θα πρέπει να γίνουν σε ό,τι αφορά την ευαισθητοποίηση. Ένα παράδειγμα. Πήγαμε και στην Amazon για να αγοράσουμε την κούκλα. Ή την Amazon ή σε κάποιο άλλο κατάστημα. Κοιτώντα τα σχόλια τι κριτικέ των γονέων. Γιατί παραπονιούνται οι γονεί, Ότι την κούκλα δεν καταλάβαινε τον παιδικό τρόπο μιλήσει των παιδιών του. όλα τα υπόλοιπα δεν του ενδιαφέραν. Βαθιά ανοιχτωμένοι. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε τα πιο πολλά εργαλεία στο GPDR και στη privacy, αλλά κάποιες από τις νομοθεσίες που ισχύουν ακόμα εξακολουθούν να είναι παροχημένες, θεωρούμε. Για παράδειγμα, οι αρχέ για την προστασία των για την προστασία των, της ασφάλειας των παιδιών. Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας για την Google αυτή, για παράδειγμα. Η νομοθεσία έχει να κάνει πιο πολύ με τον άμεσο Και τον άμεσο κίνδυνο. Μπορεί το παιδί να πάθει κάτι άμα φάει την κούκλα, για παράδειγμα, άμα φάει η τρίχα τη κούκλα. Αλλά υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι πέρα από αυτού του άμεσου κινδύνου. Ευχαριστώ πολύ και ο κύριο Νέμετσε. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι η πρόκληση ε, των χρόνων ε, τώρα είναι ε, να κάνουμε πιο εύκολη την δουλειά για τους μεμονωμένους ανθρώπους. Ε, δηλαδή θα πρέπει να δούμε ε, με ποιο τρόπο μπορούμε να βοηθήσουμε την ε, τεχνολογία επιβολής με τον τρόπο δηλαδή με τον οποίο μπορούν τα ίδια τα άτομα να ελέγξουν για τα δεδομένα τους έτσι ώστε ε, και οι επόπτες αλλά και οι μεμονωμένοι ε, πολίτες να έχουν την δυνατότητα να ελέγξουν ε, αυτά τα, αυτές τις νέες δυνατότητες. Έχουμε τη δυνατότητα να είμαστε high-tech, έχουμε την δυνατότητα να είμαστε ε, σε θέση να, ε, να χρηματοδοτήσουμε τα DPAs έτσι ώστε να ε, κάνουν ας πούμε κάποια χειρίδια. αλλά ίσως το πιο καλό θα ήταν στο μέλλον να έχουμε μία εφαρμογή, μία application από τα DPAs έτσι ώστε να μπορέσουμε να φτάσουμε φτάσουμε σε περισσότερο κόσμο και τα χρήματά μας να πιάσουν τόπο. Ε, tech for law είναι το ε, καινούριο μότο ας πούμε, το καινούριο σλόγγαν. Ε, κάτι άλλο, οι αρχές ε, προστασίας ε, των δεδομένων αλλά και κάποιες άλλες οργανώσεις προστασίας καταναλωτών και τα λοιπά θα πρέπει εκ των πραγμάτων εξοφίτσιο να μπορούν να παρεμβαίνουν σε τέτοιες περιπτώσεις παραβίασης δεδομένων τελευταίες παρατηρήσεις τα big data έρχονται στην Ευρώπη. Ε, είναι λάθος να λέμε ότι θα χάσουμε τα δεδομένα και τα λοιπά. Μα δέστε τις, ε, τα στατιστικά των ε, μεγάλων αποθηκών ας πούμε big data. Βλέπετε ότι πολλές αμερικανικές εταιρείες οικοδομούν τα δικά τους κέντρα αποθήκευσης big data στην Ευρώπη. Γιατί, μα γιατί μας εμπιστεύονται ε, ξέρετε ότι η Apple είναι η πιο, ε, είναι η πιο ε, μεγάλη εταιρεία όσον αφορά τέτοιου είδους θέματα και διαλέγει παρόλα αυτά να έρχεται στην Ευρώπη. Απ' την άλλη πλευρά και κάτι άλλο που θέλω να πω. Όποιος ας πούμε, τι να σας πω, τα big data ε, μας δίνει και την ε, δυνατότητα να αναγνωρίσουμε ε, κάποιες κατηγορίες ανθρώπων και να τις αποκλείσουμε από κάποια πράγματα. Αυτό το χρησιμοποιούν ή μπορούν να το χρησιμοποιήσουν και οι αστυνομικές αρχές. Υπάρχει βέβαια ο κίνδυνος να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα αυτά έτσι ώστε να πεις ότι ε, δεν ε, ε, ότι ας πούμε θέλω να νοικιάσω ένα σπίτι αλλά δεν θέλω να είναι λευκός, δεν θέλω να είναι μαύρος, δεν θέλω να είναι μουσουλμάνος ή οτιδήποτε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε ποιους πόρους βάζουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και επίσης πρέπει να είμαστε και αισιόδοξοι. 4% το μεγαλύτερο πρόστιμο το οποίο αναφέρεται στον κανονισμό. Πάντως πιστεύω ότι θα αναπτυχθούν μοντέλα τα οποία ε, θα διασφαλίζουν εξ αρχής την συμμόρφωση. Γιατί, γιατί ε, το πρόστιμο είναι ψηλό και επομένως ε, θα το σκέφτονται και θα θέλουν να συμμορφούνται εξ αρχής. Σας ευχαριστώ όλους πολύ, ευχαριστώ τους ομιλητές μας, ευχαριστώ που απαντήσατε στις ερωτήσεις των βουλευτών. Ευχαριστώ που μας δημιουργήσατε αυτή την τόσο πλήρη εικόνα για την όλη κατάσταση. Περνάμε ευθύ αμέσω στο δεύτερο γύρο, στο δεύτερο πάνελ. Μικρή αλλαγή φρουράς για τους πανελίστες και προσκαλώ τους ομιλητές της δεύτερης συζήτησης να καθίσουν δίπλα μου. Okay, everybody. We are resuming our... Συνάδελφοι, συνεχίζουμε. Το δεύτερο μέρος της συζήτησης έχει να κάνει με τις συλλογές, με τη συλλογή μεγάλων δεδομένων από τι διοικητικέ αρχές και γενικώ στο δημόσιο τομέα. Θα ακούσουμε και με κυβερνητικέ οργανώσεις για τη χρήση των μεγάλων δεδομένων και επίση τις εκπροσώπου των δημόσιων αρχών. Ο λόγος πρώτα στον κύριο Ρίβο Ράιτμαν, ο οποίο είναι γενικός υποδιευθυντής της ETCB, της ε, αρχής ε, της εφορίας και τελωνίων της Εστονίας. Θα μας παρουσιάσει την προοπτική της δημόσια Δίκησης. Έχετε 10 λεπτά. Ευχαριστώ. Είναι μεγάλη μου τιμή ε, για να παρουσιάσω το πώς συλλέγει φόρους η Δημόσια Αρχή της Εστονίας και πώς χρησιμοποιούμε τα μεγάλα δεδομένα. Πρώτα απ' όλα συλλογή φόρων. Αυτό το σύστημα ήδη λειτουργεί από χρόνια. Το θέμα είναι πώς συλλέγουμε πλέον τα δεδομένα και τι τα κάνουμε. Η δική μας η άποψη επί του θέματος είναι ότι η συλλογή δεδομένων για λόγους φορολογικούς θα πρέπει να λειτουργεί με δύο τρόπους. Και να σας απασχολούν εδώ δύο ζητήματα, δύο σκέλη. Πρώτα απ' όλα πώς λαμβάνουμε τα δεδομένα και δεύτερον τι τα κάνουμε. Πώς θα είναι στους επιχειρηματίες και στους πολίτες δηλαδή το όλο θέμα των δεδομένων. Υποβολή δεδομένων. Απόψή μας είναι πως είναι πολύ απλό και αυτονόητο να υποβάλει κανείς δεδομένα όσοι κρατούν βιβλία, πολίτες, επιχειρηματίες. Εν γέννη, νομίζω γνωρίζουν πώς να υποβάλουν δεδομένα. Θα πρέπει να προσφέρεται βέβαια ένα λογισμικό που να διευκολύνει την τήρηση βιβλίων και κάθε είδου ηλεκτρονικό μέσο. Τώρα για τον τρόπο που χρησιμοποιούνται τα δεδομένα στην υποβολή ηλεκτρονικών δηλώσεων και πώς εμεί φέρνουμε σπέρα τα καθήκοντά μα. Η μόνη απαραίτητη χρήση των δεδομένων για το κράτος και την εφορία είναι η φορολογική. Δεν υπάρχει λόγος να έχουμε περισσότερα δεδομένα από τα φορολογικά. Ιδανικά, τα δεδομένα θα έπρεπε να συλλέγονται ε, στο διαδίκτυο επιγραμμικά χωρίς καμία παρέμβαση. Και η δήλωση των εσόδων και η υποβολή του ποσού του φόρου θα πρέπει να γίνεται αυτομάτως. Χωρίς οι πολίτες να χρειάζεται να πάνε παραπέρα, να κάνουν κάτι παραπάνω. Δηλαδή, τα χρήματα που αυτή τη στιγμή ξοδεύουν οι επιχειρηματίε για την καταγραφή των φόρων του θα πρέπει να μένουν στι επιχειρήσει. Σε μικρέ χώρε όπω η Ιστονία, το κόστος της υποβολής φορολογικής δήλωσης είναι πάνω από 100.000 είναι πάνω από 100 εκατομμύρια ευρώ. Και τα χρήματα αυτά θα έπρεπε να παραμένουν στι εταιρείε για να επενδύουν. Δηλαδή και για τον υπολογισμό της επιστροφής του φόρου και για τον υπολογισμό γενικώ ε, του ποσού που πρέπει να καταβάλει κανείς, όλα αυτά θα πρέπει να υπολογίζονται αυτόματα. Η Εστονία ήδη έχει αναλάβει σοβαρή δράση και το 2018 όλα αυτά τα συστήματα θα ευθυγραμμιστούν και θα χρησιμοποιούνται ήδη εθελοντικά. Στόχος μας να μην συλλέγονται προβολικά πολλά δεδομένα. Δεν χρειαζόμαστε κάποια σούπερ βάση δεδομένων, δεν θέλουμε να τηρούμε τα δεδομένα ε, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απλώς θέλουμε τα απαραίτητα δεδομένα για να μπορούμε να υπολογίσουμε σωστά το φόρο. Αυτό είναι ένα παράδειγμα για το πώς θα μπορούσαν να χρησιμοποιούνται online τα λογισμικά για την υποβολή προλογικής δήρωσης. Εδώ έχουμε μια, ένα παράδειγμα συνεργασίας με τράπεζες. Και ένας επιχειρηματίας που θα θέλει να πληρώσει τους πόρους μας αυτής της εφαρμογή του online banking θα μπορούσε να υποβάλει απευθείας με τη φορολογική του δήλωση στην εφορία. Θα υπολογιζόταν ε, το ποσό του φόρου και ο φόρος να πληρώνεται απευθεία. Δεν θα χρειαζόταν να συμπληρώσει κανένα επιπλέον έντυπο. Μιλάμε δηλαδή για μια μεταφορά ποσού, όπως είναι τη μεταφορά των ε, μισθών ε, με έμβασμα στο τραπεζικό λογαριασμό. Το πιο σημαντικό πάντως είναι τι τα κάνουμε αυτά τα δεδομένα. Τα δεδομένα που συλλέγουμε δεν ανήκουν στο κράτος. Ανήκουν στους επιχειρηματίες και στους πολίτες. Σε αυτούς που τα υπέβαλαν. Πρέπει λοιπόν να δίνουμε την απαραίτητη αξία τους σε αυτά τα δεδομένα και να τα επιστρέφουμε και στους κατόχους τους. Το θέμα είναι πώς τα ε, υποβάλλουμε ξανά και πώς τα επιστρέφουμε στους κατόχους. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε προσωπικά στατιστικά στοιχεία βάσει αυτών των δεδομένων να ξέρω ας πούμε ποιος είναι ο μέσος όρος των μισθών στην κομιτεία ή την επαρχία όπου κατοικώ, πόσο κερδίζει ο κόσμος, πώς μπορώ να βρω, τι δουλειά μπορώ να βρω βάσει των προσόντων μου. Βάσει όλων των δεδομένο που απαιτεί το κράτος θα έπρεπε οι πολίτε να μπορούν να έχουν πρόσβαση και σε αυτέ τι πληροφορίε όπω το κράτο, αυτή τη στιγμή ε, Μάλλον, επίση οι επιχειρηματίε είναι καλό να γνωρίζουν πώ έχει το οικονομικό περιβάλλον, ποιο είναι ο κύκλο εργασιών κάποιων εταιριών, εάν είναι ανταγωνιστικοί στι εταιρείε του ή όχι. Όλε αυτέ είναι οι αποφάσει που μπορεί να πάρει κανεί όταν έχει τα απαραίτητα δεδομένα. Και υπάρχει σε αυτά πρόσβαση. Ένα άλλο σημαντικό παράγοντας είναι η διαχείριση του κινδύνου. Οι φορολογικέ αρχέ της ευρωπαϊκής χώρες πραγματοποιούν μελέτες αντικτύπου για να δουν ποιο προσπαθεί να αποφύγει φόρους και να φοροδιαφύγει. Τα δεδομένα αυτά τηρούνται από τους αρμόδιους φορείς και τις αρχές και αυτέ οι πληροφορίε μεταφέρονται αλλού μόνο όταν υπάρχει κίνδυνο επιβολή κυρώσεων. Εμεί πιστεύουμε ότι αυτά τα δεδομένα θα έπρεπε να διατίθενται εφόσον χρειάζεται και προσπαθούμε μετά τι ε, πληροφορίε να τι προσφέρουμε πίσω στι επιχειρήσει αφού συμπληρωθούν, για να δουν ε, και επιχειρηματίε λόγω χάρη πώ τους βλέπει το κράτο. ποιοι είναι κίνδυνοι να μπορέσουν να ετοιμάσουν κατευθυντήρε γραμμέ για να περιορίσουν στο ελάχιστο τον κίνδυνο φοροδιαφυγή. Θα θέλαμε να έχουμε μια τέτοια υπηρεσία που οι επιχειρηματίες να βλέπουν συστημικό κίνδυνο και να μπορούν να μεγεραστούν το θέμα ε, τη συγκεκριμένη πληροφορία με άλλους επιχειρηματίες να τα δημοσιεύσουν και επιγραμμικά. Δηλαδή να πει κανείς αυτή είναι η φορολογική συντελεστέ, συνεργαστείτε μαζί μου. Τα δίνουμε λοιπόν αυτά στους άλλους επιχειρηματίες, θα μπορούσαν να τα μοιράζονται με συναδέλφους τους και εμείς Ω φορολογικέ αρχέ δεν χρειάζεται να τηρούμε πια αυτέ τι πληροφορίε, μπορούν να τι αναλάβουν στα χέρια του οι ίδιε εταιρείε. Στατιστικά δεδομένα είναι και μοίρασμα, κατανομή των πληροφοριών για όλη την Εστονία, αλλά θα μπορούσε να συμβαίνει αυτό και σε όλη την Ευρώπη. Έτσι θα είχαμε μια καλή βάση για συγκρίσει και για όλους τους επιχειρηματίες στην Ολλανδία λόγω χάρη, την Εστονία και ούτω καθεξής. Πιστεύω ότι ένα τέτοιο σύστημα θα ήταν πραγματικά εύκολο να δημιουργηθεί. Οι επιχειρηματίε μπορούν να αναλάβουν τη διαχείρισή του και δεν μιλάμε για δημόσια δεδομένα που τα δημοσιεύει το κράτο, αλλά ίδιε εταιρείε και οι ενδιαφερόμενοι. Ευχαριστώ για την προσοχή σα. Επίση, να θυμίσω ότι η δική μα δουλειά δεν είναι υποπτία των επιχειρηματιών. Δεν θέλουμε να του αστυνομεύουμε για να είμαστε χωροφύλακε, αλλά να του προσφέρουμε consulting. Ευχαριστούμε. Α προχωρήσουμε τώρα στο δεύτερο μιλητή, στον κύριο Ραούλ Ζάβημα, από την Αστυνομική Αστυνομία και Συνοριοφυλακή. Από την Εστονική Αστυνομία λοιπόν και Συνοριοφυλακή. Σας ευχαριστώ πολύ. Honorable. Αξιότιμοι βουλευτέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίε και κύριοι. Θα σα περιγράψω πώ χρησιμοποιείται τα big data στην, ε, ε στον νόμο σε ό,τι αφορά τη συνοριοφυλακή και την αστυνομία τη Εστονία. Και μια και έχουμε και διερμηνία, να μιλήσω στον Για την παρουσίασή μου τουλάχιστον. Ε, η δική μας εκτίμηση είναι ότι το big data δίνει μεγάλες ανοίγει μεγάλες δυνατότητες για την αστυνομική υπηρεσία, για την αστυνομία. Αλλά υπάρχουν και περιορισμοί, τα big data, όπως όλα τα δεδομένα που μας χορηγούνται. Για να πετύχουμε τους δικούς μας στόχους, πρέπει να πούμε ότι έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Υπαγόμαστε στο Υπουργείο Δικαιοσύνη, αλλά σύμφωνα με το δίκαιο τη Εστονίας, ο εισαγγελέα είναι ο υπεύθυνο για την εξαγωγή των ερευνών. Όταν δεν χρησιμοποιούμε τα δεδομένα, τα χρησιμοποιούμε πάντα με την συνένεση του εισαγγελέα. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν η χρήση των δεδομένων και η αξιοποίηση των δεδομένων ακολουθεί τις αρχές αυτές και σε καμία περίπτωση δεν ε, μπορεί να υπάρχει οποιαδήποτε διαδικασία παρακολούθησης χωρίς να έχει ανοίξει μια επίσημη ε, έρευνα. Υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις ασφαλώς, αλλά γενικά είναι πάρα πολύ επακριβής και αυστηρή η κανόνα στη σχετική για τη χρήση των δεδομένων από τις αρχές επιβολής του νόμου στην Εστονία. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα δεδομένα αυτά τα οποία μας επιτρέπει η νομοθεσία της Εστονίας να χρησιμοποιήσουμε. Χρησιμοποιείται λοιπόν τα δεδομένα για να αναλυθεί η κατάσταση στο κλιματικό τοπίο, για να γίνουν προγνώσεις και προβλέψεις για τις ενδεχόμενες εξελίξεις. Έχουμε και ένα σύστημα φύλαξη των δεδομένων. Πρόκειται για ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει διάφορα στατιστικά πακέτα από διάφορες βάσεις δεδομένων και σκοπός και στόχος του συστήματος είναι να αξιολογηθεί η κατάσταση σε ό,τι αφορά την εκτέλεση, των, την επιβολή του νόμου σε διάφορες κοινότητες, σε διάφορες περιοχές και περιφέρειες της Εστονίας. Αλλά χρησιμοποιούμε αυτό το σύστημα πληροφοριών για να κάνουμε και προβλέψεις για το πού θα πρέπει να καταβληθούν πιο μεγάλες προσπάθειες ή που θα πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε ε, πιο συντονισμένες προσπάθειες για την αποτροπή και πρόληψη του εγκλήματο. Φυσικά, προκειμένου να διαχειριστούμε τα δεδομένα μας, τους πόρους μας, πρέπει να χρησιμοποιούμε διάφορα δεδομένα και πολλά τέτοια δεδομένα είναι ανωνυμοποιημένα. Κάτι άλλο που είναι επίση πάρα πολύ σημαντικό είναι η ποιότητα των δεδομένων. Έχουμε δημιουργήσει ένα σύστημα ποιοτικών δεδομένων. Θέλουμε να είναι αξιόπιστα, βλέπετε, τα στοιχεία αυτά, τα δεδομένα αυτά. Αυτό είναι ο σκοπό του συστήματο. Φυσικά, ακόμα και οι αρχέ επιβολή του νόμου κάνουν ε, λάθη σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά δημιουργήσαμε ένα σύστημα το οποίο μας βοηθά να αποτρέπουμε τέτοια σφάλματα ακριβώς. Χρησιμοποιούμε λοιπόν τα big data για την ανάλυση των δραστηριοτήτων των αστυνομικών οχημάτων. Από το 2004 και μετά έχουμε ένα σύστημα GPS σε 500 αστυνομικά οχήματα. Έχουμε και κλειδαριές για την ταχύτητα, για την θέση των αστυνομικών οχημάτων αυτών. Έχουμε λοιπόν όλες τις πληροφορίες για όλες τις κινήσεις όλων των αστυνομικών οχημάτων. Ξέρουμε ποιο όχημα, ποιο όχημα βρίσκεται πού σε ποια πόλη και ξέρουμε ποιε είναι οι περιοχέ οι οποίε χρειάζονται πιο πολλά περιπολικά και πιο πολλέ περιπολίε. Στην αρχή, ασφαλώ, να ξεκίνησε το σύστημα αυτό, αστυνομικοί ήταν και κάπως ανήσυχοι. Φοβούντουσαν μήπως οι προϊστάμενοι τους επρόκειτο να τους παρακολουθούν. Ανά πάσα στιγμή, ως τώρα, ως τώρα, μέχρι σήμερα. Έχουν καταλάβει ότι ο σκοπός του συστήματος αυτού ήταν να βελτιωθούν τα συστήματα. Αυτό το σύστημα λοιπόν της ηλεκτρονικής αστυνόμευσης συνεπάγεται επίσης ότι τα αστυνομικά αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα όλα τους και με υπολογιστές. Και για την προστασία των δεδομένων, φροντίζουμε τα δεδομένα αυτά να μην φυλάσσονται ποτέ στα οχήματα, στα υπολογιστές των οχημάτων. Πάντα σε ένα κεντρικό σερβερ φυλάσσονται τα δεδομένα αυτά. Τα ανωνυμοποιημένα αυτά μεγάλα πακέτα δεδομένων χρησιμοποιούνται και σε συνεργασία με τα πανεπιστήμια και με μια εταιρεία που ονομάζεται Κούπαθ και η οποία μας χορηγεί αξιόπιστα δεδομένα για τις τηλεφωνικές κλήσεις από τις συμφωνίες που συνάπτουν με τους ε, καταναλωτές επιτρέπεται η παροχή στην αστυνομία τέτοιων ανωνυμοποιημένων στοιχείων. Και από ένα παράδειγμα από το 2011 μπορείτε να δείτε τον Ιούλιο του 2011 και τον Αύγουστο σε μία μικρή πόλη Άψαλα στην Εσθονία τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιήθηκαν πολύ πιο εντατικά, πολύ πιο πολύ από ό,τι συνήθως. Και βλέπουμε λοιπόν πόσα άτομα ζουν στην πόλη αυτή, πόσοι άλλοι κάτοικοι εκτό τη περιοχή αυτή χρησιμοποίησαν τηλέφωνα στη συγκεκριμένη περιοχή, πόσοι αλλοδαποί χρησιμοποίησαν τηλέφωνα και όλα αυτά τα δεδομένα λοιπόν τα συλλέγουμε και ξεκινάμε να προγραμματίσουμε την επόμενη φάση. Γιατί προέκυψε ότι διεξαγόταν ένα φεστιβάλ στην συγκεκριμένη κόμμα και έτσι ε, προβλέψαμε πόσα αστυνομικά οχήματα θα χρειαζόντουσαν για την περιπολία κτλ. Τα δεδομένα αυτά τα χορήγησε η εταιρεία που σας είπα σύμφωνα με τους όρους και τις συνθήκες που προβλέπονται στα συμβόλαια της εταιρεία. Μας ενδιαφέρει και ένα νέο project για την κινητή χρήση δεδομένων. Πρόκειται λοιπόν για ένα project το οποίο θα προγραμματίσει την υποδομή για την χρήση μεγάλων δεδομένων σε πανεπιστήματα, σε υπουργεία, σε αρχές επιβολής του νόμου και σκοπός είναι όλα τα δεδομένα τα οποία χρειάζονται, τα οποία χρησιμοποιούνται, να περάσουν από τη διαδικασία ανωνυμοποίησης. Επίσης, έχουμε και ένα project για να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα για το έγκλημα και για την ασφάλεια. Θέλουμε λοιπόν να παρέχουμε διάφορα δεδομένα τέτοια στην κοινωνία. Και πάλι μιλάμε για ανωνυμοποιημένα δεδομένα για διάφορα εγκλήματα. Και όλα αυτά θέλουμε να τα διαθέτουμε στην ιστοσελίδα μας. Στο μέλλον, δε. Θέλουμε να τα επεξηγούμε αυτά και με, μέσω ενός διαγράμματος. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους να χρησιμοποιούν αυτά τα δεδομένα στις ιστοσελίδες μας συνολικά θα λέγαμε ότι έχουμε όλες τις σχετικές νομοθεσίες ε, και φυσικά η αστυνομία πάντα λαμβάνει υπόψη ε, όλες αυτές τις νομοθεσίες και έχουμε και τους ε, αρμοδίους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στις υπηρεσίες μας. Υπάρχει μια σχετική υπηρεσία, ένα σχετικό γραφείο. Έχουμε ε, διαδικασίες e-learning για όλους τους αξιωματούχους της αστυνομία και των λοιπόν υπηρεσιών και θέλουμε και εξασφαλίζουμε όλοι να γνωρίζουν ποιοι είναι οι κανόνες για την προστασία των δεδομένων. Έχουμε δε και εσωτερικέ τέτοιες ε, μονάδες οι οποίες είναι υπεύθυνε για την εντοπισμό τέτοιων καταχρήσεων από αστυνομικούς. Και είχαμε τέτοιες περιπτώσεις. Έχουν προσαχθεί στο δικαστήριο πλέον οι περιπτώσεις αυτές. Έχουμε λοιπόν και ένα κέντρο τεχνικής ε, ασφάλειας και ανάπτυξης ε, τέτοιων μέτρων. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την προσοχή σας και θα ήθελα να κλείσω λέγοντας ότι ξέρουμε τι είναι τα big data, αλλά εμείς στην αστυνομία θέλουμε να προστατεύουμε όλα τα στοιχεία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ, λέει και ο Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε για τις παρουσιάσεις αυτές. Και τώρα, ο ομιλητής, η κυρία Φρεντερίκε Καλτάουνερ, η οποία οργάνωται για την Privacy International, μία ΜΚΟ, και θα μας πει τι γίνεται στις δημόσιες αρχές ό,τι αφορά την προστασία Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με καλέσατε να μιλήσω εδώ. Εγώ εργάζομαι για την Privacy International. Είμαστε φιλανθρωπική οργάνωση με βάση το ε, Λονδίνο και ασχολούμαστε με επίλυση διαφορών ε, με επιχειρήσεις κυρίως όσον αφορά ανθρώπινα δικαιώματα. Είναι αδύνατον ε, να ζήσει κανείς στη σύγχρονη ζωή χωρίς να παραγάγει πολλά προσωπικά δεδομένα. Ε, πιστεύουμε ότι, ε, ε, συγγνώμη, στη ζωή που ζούμε, από το να πιούμε ένα καφέ μέχρι να κάνουμε μια αγορά, μπαίνουμε στην διαδικασία να δημιουργούμε δεδομένα. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να καταλάβουμε τι σημαίνει big data. Ε, πρώτα απ' όλα ε, με, την, ε, με τον όρο big data καθορίζουμε μια, ένα τεχνικό, μια τεχνική συλλογή στοιχείων. Όμως τα big data είναι και η υπεποίθηση ότι, υπάρχει, ότι δίνουν την δυνατότητα δυνατότητα να μας δώσουν στοιχεία τα οποία δεν μπορούσαμε να έχουμε πριν. Ε, ε, αυτό αναφέρεται και ότι μπορεί να επηρεάσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό μπορεί να χρησιμεύσει, ας πούμε, και ισχύει για τα κοινωνικά δίκτυα κτλ η τεχνολογία μπορεί να τροποποιήσει με πολύ, με πολύ σημαντικό τρόπο τα big data. Ε, εδώ θα σας δείξω μια μελέτη φοιτητών σχετικά με το τι σημαίνει ακριβώς big data. Εάν ας πούμε ε, τα αρχεία της ε, Στάζη, τα, βάζαμε στη σειρά, θα δημιουργόταν αυτός ο διάδρομος κατά κάποιο τρόπο. Εδώ ε, βλέπετε την διασύνδεση ανάμεσα σε τεχνολογία και δεδομένα με πολύ πρόσφατα παραδείγματα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ε, αναφερόμενο, ένα άρθρο αναφέρθηκε στις ε, ε, εκλογές στην Αμερική και αναφερόταν ότι μια εταιρεία βρετανική δημιούργησε κάποια ψυχομετρικά προφίλ ε, τα οποία μπορούσε να χρησιμοποιήσει, ε, τα οποία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ε, και τα έδωσε στον ρεπουμπλικανό υποψήφιο για ολόκληρη την Αμερική και θεώρησε ότι με, την, ότι με αυτόν τον τρόπο έδινε δυνατότητα δημιουργίας 5.000 προφίλ. Ε, όμως ε, δεν είναι ε, σωστό αυτό, δεν είναι δυνατόν δηλαδή μια μεγάλη εταιρεία marketing ή ένα είδος big data ότι μπορούν υποτίθεται να επηρεάσουν εκλογές και δεν υπάρχει κανένα αποδεικτικό στοιχείο ότι αυτός ο τρόπος στόχευσης λειτουργήσε. Ταυτόχρονα ναι. υπάρχουν παραδείγματα τα οποία απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα big data μπορούν να παραβιάσουν τα θεμελιώδη δικαιώματα. Ας πούμε σε περίπτωση ε, ε, ε, πολύ ευαίσθητων πληροφοριών σχετικά με την σεξουαλική ζωή των ανθρώπων ε, μπορούν να ε, ε, γίνουν γνωστά. Δηλαδή ακόμα και οι καταναλωτές οι οποίοι είναι πολύ προστεκτικοί στα στοιχεία τα οποία δίνουν στα, στα μέσα δικτύωσης κοινωνικής μπορεί να πέσουν στην παγίδα αυτή. Βεβαίως εδώ το ερώτημα που προκύπτει είναι ο διαχωρισμός ανάμεσα σε προσωπικά και μη προσωπικά δεδομένα. Το παράδειγμα αυτό δίνει, δείχνει επίσης ότι οι προβλέψεις ενδεχομένως ε, δεν είναι σωστές ε, ή είναι σαφώς μεροληπτικές. Ε, αυτή, αυτού του είδους η μεροληψία μπορεί να οδηγήσει ε, σε διακριτική μεταχείριση ε, και αυτό μπορεί να έχει πολύ κακές επιπτώσεις σε περίπτωση ας πούμε ελέγχου ε, για προαγωγή ή για πρόσληψη ή για λόγους αστυνομικής επιβολής. Βεβαίως το θέμα είναι ότι πολύ συχνά οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν καν ότι ταξινομούνται ή ότι το προφίλ τους ενημερώνεται. Βεβαίω, εάν εγώ δεν ξέρω ότι κάποιος κάνει το προφίλ μου ε, δεν μπορώ να έχω και πληροφορίες για τον τρόπο με τον οποίο το προφίλ μου καταρτίζεται. Στην οργάνωσή μας ε, θέλουμε να πούμε ε, ότι η πληροφόρηση, η πληροφορία δίνει εξουσία και η εξουσία ε, ε, διαφθείρει. Αλλά βεβαίως το σημαντικό είναι αυτό το ε, ψήγμα, αυτό το τμήμα γνώσης το οποίο μπορεί να έχει ο, κανέν, ο καθένας είτε πρόκειται για, ασκή, για άσκηση επιβολής του νόμου είτε πρόκειται για στοιχεία τα οποία οπωσδήποτε οδηγούν σε παραβίαση των ανθρωπίνων και θεμελιωδών δικαιωμάτων. Ε, εμείς θεωρούμε ότι καμία αρχή δεν μπορεί να έχει αυτήν την ε, δικαιοδοσία στα χέρια της και αυτό συμβαίνει στις ΗΠΑ τώρα τελευταία. Ε, ένα στοιχείο το οποίο ε, αξίζει την προσοχή μας ε, είναι ότι πέρα από τα δεδομένα τα οποία κινούνται ή διακινούνται μέσω των ε, κοινωνικών δικτύων υπάρχουν και άλλα στοιχεία. Προχωρούμε λοιπόν έχοντας ε, κατά νου πιο προχωρημένες καταστάσεις, ε, οι οποίες μπορούν να αφορούν ε, ακόμα και την κίνηση σε εσωτερικούς χώρους ή επιλογές απολύτως προσωπικές. προσωπικές. Επίσης, όσον αφορά την επιβολή του νόμου, δημιουργούνται όλο και περισσότερο εργαλεία επιτήρησης, εργαλεία αστυνόμευσης κτλ. Όλα αυτά τα εργαλεία ε, ε, βρίσκονται ε, στο χαστρό για τους ίδιους λόγους που ανέφερα και προηγουμένως, γιατί οδηγούν σε παράβαση, παραβίαση του προσωπικού χώρου καθώς και μπορούν να οδηγήσουν ακόμα και σε μεροληπτικές και διακριτικές συμπεριφορές. Στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε γνώση του ότι πολύ συχνά ε, η αστυνομία χρησιμοποιεί εργαλεία τα οποία έχουν ε, δημιουργηθεί για τον ιδιωτικό τομέα, ή την ιδιωτική ε, σφαίρα. Όσον αφορά την, την προγνωστική ας πούμε στην αστυνομία, ξέρουμε ότι υπάρχουν πολλές και διαφορετικές μεθοδολογίες οι οποίες μπορεί να αντιτίθενται, μπορεί να βασίζονται μάλλον σε αστυνομικά στοιχεία ή σε στοιχεία τα οποία έχει μαζέψει ε, η κυβέρνηση, τα οποία βρίσκονται ε, και έχουν συλλεγεί από κοινωνικά μέσα δικτύωσης ε, κλπ. σε σχέση με αυτά που έλεγε και ο συνάδελφο από την Εστονία, εγώ αναφέρομαι περισσότερο ε, σε πιο ε, αδρές ε, περιπτώσεις. Ας πούμε, στην Καλιφόρνια χρησιμοποιείται ένα είδος λογισμικού το οποίο έχει την δυνατότητα να διασταυρώσει πάρα πολλά στοιχεία από κτηματολόγια μέχρι στοιχεία ταυτότητας αγορών κτλ. Mm. Εδώ πάλι υπάρχει ένα πρόβλημα διαχωρισμού ανάμεσα στον μύθο και την πραγματικότητα. Ε, υπάρχει μια τάση να έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στις αναλυτικές μεθόδους ε, και στα ε, big data. Ε, τα εγχειρίδια της αστυνομίας όμως αναφέρουν όλο και περισσότερο το γεγονός ότι τα προηγουμένα μαθηματικά και η δύναμη των υπολογιστών δεν είναι από μόνα τους αρκετά έτσι ώστε να αποτρέψουν ε, το έγκλημα. Θα τελειώσω αναφερόμενοι σε ορισμένα στοιχεία τα οποία αφορούν ε, την διασύνδεση κινδύνου ή επικινδυνότητας μάλλον ε, ενός ατόμου που ενδεχομένως θα μπορούσε στο μέλλον να διαπράξει κάποιο έγκλημα. Αυτό μας απασχολεί πολύ. Ένα άλλο που μας απασχολεί είναι ε, να χρησιμοποιούνται ε, στοιχεία τα οποία είναι δημόσια ε, και δημοσίως διαθέσιμα έτσι ώστε να δημιουργούνται διασυνδέσεις οι οποίες αφορούν την προσωπική ζωή ατόμων ή, ή ομάδων ατόμων. Μια δίκαιη ανησυχία που έχουν όλοι είναι ότι δεν υπάρχουν ε, στοιχεία που να είναι τελείως πλήρη και χωρίς προκαταλήψεις ή κάποια πράγματα που είναι ιδέες που έχουν προδιαμορφωθεί. Όλα αυτά θα διέπονται από κάποια ε, λανθασμένη αρχική ιδέα και θα υπάρχει διακριτική μεταχείριση των ίδιων δεδομένων. Επόμενη διαφάνεια. Να προσθέσουμε ότι θεωρητικά όλα τα εργαλεία της αστρονομίας που επιτρέπουν τις προβλέψεις είναι λογισμικό με ε, συγκεκριμένο κάτοχο που πολλούνται σε υπηρεσίες και των ε, ιδιωτικών ε, εταιριών επιβολής της ασφάλειας. Άρα, για να ολοκληρώσω, είναι σωστή κατεύθυνση των μεγάλων δεδομένων και του συνδυασμού του με τα προσωπικά δεδομένα, όμω υπάρχουν και σοβαρότατε πτυχέ, οι οποίε πρέπει να μελετηθούν περαιτέρω ή έστω να καλυφθούν από την οδηγία για την ηλεκτρονική ασφάλεια. Λόγω χάρη ε, ότι τα δεδομένα θα πρέπει να είναι ανώνυμα ε, ότι θα πρέπει να υπάρξει διάκριση μεταξύ της συλλογής των δεδομένων και της παραγωγής δεδομένων και ότι όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με έναν τρόπο στα πλαίσια της νομοθεσίας. Σας ευχαριστούμε για αυτή την παρουσίαση και τώρα θα δώσω το λόγο στα μέλη. Στα μέλη που θέλουν να πάρουν το λόγο. Η συγγήτρια κυρία Γκόμες και όποιος άλλος θελήσει. Πρώτα απ' όλα για τις παρουσιάσεις από την, από την Εστονία, για τους φίλους μας αυτούς. Ο τρόπος που χρησιμοποιείται η τεχνολογία είναι αρκετά εντυπωσιακό. Και έδωσε καλά αποτελέσματα. Αλλά είναι και πολύ προσεκτική η τήρηση των δεδομένων, η όλη διαχείριση, γιατί καταλαβαίνω ότι μιλάμε για εφορία, φορολογικά, Οπότε την όλη σας δράση την βασίζετε στη συνένεση και φαντάζομαι στην ε, συνειδητή συνένεση των πολιτών. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό να είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για να καταπολεμήσουμε την συλλογή, την φοροδιαφυγή μάλλον, τη φοροαπάτη και άλλου είδους οργανωμένο έγκλημα, και άλλων ειδών οργανωμένο έγκλημα, αλλά η ερώτησή μου είναι έχετε πρόσβαση μόνο από μία υπηρεσία και πρέπει απλώς να είναι κανείς βέβαιος ότι θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι πληροφορίες που χρειάζονται. Πόσο τα μοιράζεστε όμως αυτά με άλλες δικτικές αρχές, με αρχές επιβολής του νόμου. Είπαμε για συγκεκριμένους σκοπούς. Αλλά ξέρω εγώ, ας πούμε ότι θέλετε να τα χρησιμοποιήσετε για καταλαμμίσεις της τρομοκρατίας. Μπορεί να αλλάξει απλώς ο τίτλος των δεδομένων. Πώς γίνεται λοιπόν στην πράξη η αλλαγή. Επίσης, κυρία Καλτόιτνα, έτσι σας λένε. Καλτόιτνα, Καλτόινερ. Μιλήσατε για τον κίνδυνο αυτά τα στοιχεία να τα πάρουν στα χέρια τους και οι ιδιωτικέ εταιρείες που πουλάνε υπηρεσίες ασφάλειας. Το θέμα είναι λοιπόν ε, πώς θα διαμορφωθεί αυτό το δίκτυο, πώς θα ελέγχουμε αυτούς τους μηχανισμούς, όμως και εσείς κύριε Σαβήμα, ξέρετε και τι συμβαίνει στο Πανεπιστήμιο του Ταρτού και μπορείτε εκεί να αναπτύξετε το κατάλληλο σύστημα παρακολούθησης. για τη συλλογή των προσωπικών δεδομένων και γενικώ την προστασία τους. Και σε όλους εσάς ήθελα να ρωτήσω το εξής η συνέπεια της συνάθρεσης δεδομένων, της συμπίλησής τους από διαφορετικά δεδομένα και πηγές. Τι ιδιαίτερες πληροφορίες εγείρει. Ε, τι ιδιαίτερες δυσκολίες εγείρει. Ζούμε σε αυτή την εποχή που δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τόσα συμβαίνουν. Πρέπει λιγάκι να προλάβουμε Τη εξέλιξη των καιρών. Ή θα πρέπει να νομοθετήσουμε να αλλάξουμε συμπεριφορά από την πλευρά των νομοθετών, των χρηστών, αλλά σαφώς η κοινή γνώμη δίνει προσοχή σε αυτό το θέμα. Και η κοινή γνώμη ξέρει ότι από αυτό επηρεάζεται η συμπεριφορά της, ε, ανάντι και κατάντι. Υπόθηκε λοιπόν ότι είναι πολλά τα καλά που μπορούμε να πετύχουμε με, τους με τα μεγάλα δεδομένα, αλλά είναι πολύ κίνδυνοι και οι περιπτώσει ε, από ιδέε προκαθορισμένε να οδηγηθούμε σε διακριτική μεταχείριση. Τέλος πάντων, να φτάσω και σε αυτή την ερώτηση την περίφημη. Για το DDPI τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων έχει συνέπειε ε, για την ε, συμπεριφορά όλων μα. Υπάρχουν κάποιοι κανόνε που του σεβόμαστε ή όχι, αλλά τι γίνεται με κάτι άλλο που μας ενδιαφέρει, με κάποιον άλλο που εδώ μα ενδιαφέρει πάρα πολύ εδώ. Η Κίνα. Δεν βλέπω να ανησυχούν ε, οι υπηρεσίε τη κυβέρνηση που δίνουν συμβάσει στι κινέζικε εταιρείε όπω η Huawei η οποία είναι ευημερία της Κίνας θα πει το όνομα. Αυτή είναι η κυριολεκτική μετάφραση του Huawei. Και μας είπαν ότι έχουν ένα κανόνα βάσει το οποίο οι κοινωνιζικές αρχές τους υποχρεώνουν να τηρούν κάθε δεδομένο που φτάνει στα χέρια τους. Ανησυχεί αυτό κανέναν. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και η κυρία Βερζιά έδωσε το λόγο και μετά θα ακούσουμε τις απαντήσεις. Για δύο λεπτά παρακαλώ το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ και τους τρεις. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Να σας ε, πω όμως και το εξής ως παρατηρήσει. Θεωρώ ότι μας μιλήσατε πάρα πολύ για τα πλεονεκτήματα και μιλώ και στους εκπροσώπους της Εστονίας σας συγκεκριμένα. Μας μιλήσατε λοιπόν πάρα πολύ για τα πλεονεκτήματα των συστημάτων που βασίζονται βασικά σε θέματα καλής θέλησης και στην ε, λογική ότι υπάρχει κεφάνεια. Κατανοητό. Μας είπατε ότι υπάρχουν και κίνδυνοι δεν μας εξηγήσατε όμως ε, πώς θα αποτραπούν οι κίνδυνοι αυτοί. Ε, εδώ λοιπόν θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή. Να προσθέσω δε και το εξή. Νομίζω ότι υπάρχει διαφορετική κουλτούρα στο ιστορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα αυτά. Αυτά που γίνονται στην Εστονία ενδεχομένως να μην γίνονταν τόσο εύκολα με τους ίδιους όρους και αλλού. Αυτό ό,τι αφορά την ιδέα σα ε, να γενικευτούν κάποια τέτοια συστήματα. Δεν γίνεται λοιπόν όλα σε όλε τι χώρε. Εγώ είμαι Γαλλίδα, ξέρετε, και έχουμε μεγάλη παράδοση στην δυσπιστία. Εντάξει, δεν είναι πάντα δικαιολογημένη αυτή η δυσπιστία. Αυτός που έχει καεί, ξέρετε, στο χείλο, φυσάει και το γιαούρτι μετά. Και νομίζω ότι υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα εξασφαλίσουμε. Πείτε μας λοιπόν ποιες είναι οι εμπειρίες που είχατε με το θέμα αυτό τώρα, γιατί αναφέρατε ότι υπάρχουν κίνδυνοι και μας παρουσιάστηκαν και συστήματα και πείτε μας λοιπόν τι πιστεύετε. Μας είπατε επίσης ε, ότι υπάρχουν κάποιοι κίνδυνοι, αλλά δεν μας προτείνατε ιδιαίτερα ε, λύσεις ε, για να αποφύγουμε τους κινδύνους αυτούς σε ό,τι αφορά για παράδειγμα το τι θα συμπληρώνονταν ενδεχομένω η νομοθεσία για, κάποια θέματα. Πείτε μας λοιπόν, γιατί θεωρώ την ευθύνη μας ως νομοθέτες να βρούμε τέτοιες λύσεις, να προσπαθήσουμε να βρούμε λύσεις για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε ακριβώς ε, τους κινδύνους αυτούς και να βελτιστοποιήσουμε τις εργασίες μας στον τομέα αυτό. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Λάνστιν. Να, πω λόγια για τη χρήση των μεγάλων δεδομένων στην φρολογία. γιατί είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον ε, αυτά που μας είπε και η Άννα από την Επιτροπή, που είναι και στην Επιτροπή, Εντάξει, Πείτε μας για το ΦΠΑ. Γιατί ο φόρος ε, ο φορολογίας δήματος είναι πιο απλή υπόθεση. Ακούσαμε και πάρα πολλά ζητήματα για απάτη στο ΦΠΑ και μας λένε ότι ο ΦΠΑ είναι και πολύ περίπλοκος. Δεν μπορεί να εφαρμοστούν διαφορές στο ΦΠΑ για διάφορου τομεί, για διάφορε περιοχέ, γιατί είναι τόσο δύσκολο να υπολογιστεί. Φρικτό. Πείτε μα λοιπόν τι γίνεται με το ΦΠΑ λίγο πιο συγκεκριμένα και κάτι άλλο. Όπω είπε και η αστυνομία και ήταν πάρα πολύ καλό που το ακούσαμε, πολύ ενδιαφέρον, ότι εργάζονται για να υπάρχουν ε, ανοιχτά δεδομένα. Τι γίνεται και με τις φορολογικές ε, αρχές, γιατί με ενδιαφέρουν ως επιστήμον τα συστήματα αυτά, τα φορολογικά αυτά συστήματα, αλλά δεν είναι δυνατόν να υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Για παράδειγμα, οι πολιτικοί σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα αυτά, ε, οι υπουργοί οικονομικών κτλ. Όχι όμω οι οικονομολόγοι που εργάζονται στον ακαδημαϊκό κόσμο και στην πανεπιστήμη. Τι γίνεται λοιπόν με τη δημόσια αυτή πρόσβαση στα δεδομένα αυτά Μέχρι πού μπορεί να φτάσει αυτή η ανοιχτή πρόσβαση σε αυτό το βουνό, τον όγκο το μεγάλο δεδομένων. Ευχαριστώ πάρα πολύ και θα ήθελα και εγώ να προσθέσω τέλος ένα-δύο σχόλια και μια-δύο ερωτήσεις και να δώσω μετά το λόγο και στους ομιλητές για να απαντήσουν. Άκουσα και είδα ότι υπάρχουν διαφορές λίγο μεταξύ των όσων μας είπε η κυρία Σάβημα και αυτά που μας παρουσίασε η κυρία Καλτόνερ για το τι γίνεται στις ΕΙΠΑ από τις αστυνομικές αρχές να χρησιμοποιούν τέτοια big data μεγάλα πακέτα δεδομένων. Κυρία Σάβημα, νομίζω ότι μας είπατε ότι εργάζεστε με τα ιστορικά σας δεδομένα για τα αυτοκίνητά σας με ανωνυμοποιημένες επίσης πληροφορίες και δεδομένα. Ενώ τα άλλα παραδείγματα βασίζονται πιο πολύ σε προσωπικά δεδομένα κάποιων συγκεκριμένων υπόπτων. Και νομίζω ότι υπάρχει και μια ευκαιρία εδώ να διαπιστώσουμε μια κάποια κατεύθυνση η οποία ενδεχομένω να είναι και η σωστή και η ενδεδειγμένη. Πείτε μας λοιπόν και οι δύο κάτι παραπάνω. Μήπως υπάρχει και κάποια... κάποιος απότερος στόχος πίσω από τις διαφορετικές αυτές προσεγγίσεις. Κάτι άλλο. ένα πιο αφηρημένο, αν θέλετε, παράδειγμα, το οποίο ωστόσο θεωρώ ότι καταδεικνύει και ένα τμήμα της συζήτηση το οποίο αφορά τα όρια, τα ηθικά, τα διοντολογικά όρια. Μπορεί να υπάρχει ένας αλγόριθμος ε, μεγάλων δεδομένων, αναφέρεται, βάσει δεδομένων που συλλέγονται και να καταλήξει το συμπέρασμα ότι οι κοκκινομάλιδε, για παράδειγμα, είναι πιο ε, πιθανόν να διαπράξουν έγκλημα σε σχέση με του υπόλοιπους. Ή δεν ξέρω, μπορεί να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι μπορεί να είναι πιο πιθανό να προβούν σε απάτη, φοροαπάτη. Πολλά από τα χαρακτηριστικά αυτά ενδεχομένω να προκύψουν ως δείκτες από τους αλγοριθμούς αυτούς δείκτες συγκεκριμένων συμπεριφορών, παρά το γεγονός ότι τέτοιοι δείκτες δεν συνδέονται άμεσα και με προφανή τρόπο με οποιαδήποτε εγκληματική δραστηριότητα. Πιστεύετε λοιπόν ότι υπάρχει ένα σημείο στο οποίο τέτοια συμπεράσματα ναι μεν μπορεί να ισχύουν σε επίπεδο βάση δεδομένων αλλά δεν θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις έρευνες. Γιατί πολύ απλά θα βάλουμε ένα όριο και θα πούμε ότι ως εδώ και μη παρέχει. Δεν θα κάνουμε διαφορετική μετακρατική μεταχείριση κάποιων ανθρώπων επειδή έχουν διαφορετικό χρώμα μαλλιών. Όσο και να στέκουν τα στοιχεία. Υπάρχει λοιπόν κάποιο τέτοιο όριο. Έχετε βάλει εσείς κάπου ένα τέτοιο όριο. Και με τις κουβέντες αυτές λοιπόν θα ήθελα να ολοκληρώσω και να σας δώσω το λόγο για να απαντήσετε σε 4-5 λεπτά. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Ράιτμαν. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν μπορώ να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω με τη σειρά που τέθηκαν. Πρώτα όμως, για το πώ μοιραζόμαστε τι πληροφορίε μεταξύ των διαφορετικών υπηρεσιών. Ναι, το κάνουμε, αλλά αυστηρό απόρριτα, εμπιστευτικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πρέπει να να εξασφαλίσουμε την προστασία όλων αυτών των πληροφοριών. Πρέπει να ξέρουμε αυτό που θα πάρει τι πληροφορίε, γιατί ακριβώ θα τι χρησιμοποιήσει, ποιο είναι ο σκοπό του. Εάν δεν υπάρχει ένα πραγματικό συγκεκριμένο σκοπό, ο οποίο να είναι καταγεγραμμένο επισήμω, δεν παίρνουν τίποτα. Αυτό είναι σημαντικό. Και έχουμε ένα νόμο που στην Εστονία που λέει ότι πρέπει να μειωθεί το διοικητικό άχθο. Δηλαδή, αν κάποιο ήδη στέλνει πληροφορίε προ το κράτο, τότε μια άλλη υπηρεσία δεν μπορεί να ζητάει την ίδια πληροφορία δεύτερη φορά. Άρα, ε, εμέσω πλησαφώ αποδέχεται κανεί το μοίρασμα των πληροφοριών. Βεβαίω, έχει κανεί το δικαίωμα να ζητήσει από την άλλη υπηρεσία την πληροφορία, όμω εκεί σταματάει η κατανομή. Δηλαδή, ε, ε, από τη στιγμή που ε, καταλαβαίνει κανεί γιατί ε, δέχεται το μοίρασμα των πληροφοριών. Πρέπει να υπάρχει αποστολή μόνο των απαραίτητων πληροφοριών. Πάντως, στη βάση των δεδομένων είναι ξεχωριστά οι πληροφορίε στην κάθε υπηρεσία. Δεν μπορεί δηλαδή να μπει, κανείς να μπει σε ένα κεντρικό ιστότοπο και να δει τα πάντα. Αυτό είναι πρακτικά αδύνατο. Για το θέμα της εμπιστοσύνη. Βεβαίω υπάρχουν διαφορές στην οτροπία, πολιτιστικές διαφορές. Όμως αυτό ακριβώς θα έπρεπε να κάνει ένα κράτος για να χτίζει σχέσεις εμπιστοσύνη. Δηλαδή να συλλέγουμε δεδομένα ανθρώπων που μας εμπιστεύονται και να τους δείχνουμε ότι μπορούμε να τους ε, προστατεύσουμε. Από νομικής πλευράς, από νομοθετικής, από φορολογικής. Στην Εστονία τα πράγματα είναι σχετικά απλά, διότι ο κόσμος μας εμπιστεύεται όντως. Στο ηλεκτρονικό μας περιβάλλον δεν φοβούνται αλλά πρέπει να δείχνουμε στην καθημερινή ζωή ότι ναι, εμπιστευτείτε μας, δεν υπάρχει πρόβλημα. Εμπιστευτείτε μας, δεν πρόκειται να υπάρξει διαρροή. Που καμία έννοια. Και πώς το κάνουμε αυτό, έχουμε ξεχωριστές βάσεις δεδομένων, δεν χρησιμοποιούμε μια σούπερ βάση για όλα τα δεδομένα και δεν είναι τόσο πολύπλοκα τα πράγματα. Για το θέμα του ΦΠΑ. Βεβαίω είναι αρκετά περίπλοκο διότι πραγματικά είναι η απλούστερη περίπτωση που μπορεί κανεί να φοροδιαφύγει. Όμω αυτό που έχουμε δει είναι ότι πίσω από την πολύπλοκη νομοθεσία τα μικρά κομμάτια της νομοθεσίας στην τήρηση των βιβλίων γίνονται σεβαστά. Διότι ο κόσμος καταγράφεται που λέει, αγοράζει κατά λεπτός. Αυτές οι πληροφορίες τώρα. μπορούν να οδηγήσουν σε έναν αλγόριθμο για να δούμε πώς υπολογίζει κανείς τους φόρους του. Πώς συλλέγει τις πληροφορίες, τι πουλάει, τι πληροφορίες ή αγαθά. Βάσει όλων αυτών των παραμέτρων μπορεί να έχει και έναν αλγόριθμο και αυτές τις πληροφορίες να αλλάξουν. Δηλαδή, βλέπουμε το ελάχιστο ποσό από τους λογαριασμούς και υπολογίζουμε κατά μέσο όρο τον φόρο. Έτσι είναι πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Αν αλλάξει ο νόμος, το λογισμικό των εταιριών που παρέχουν το λογισμικό ακριβώ για την τήρηση των ηλεκτρονικών βιβλίων αλλάζει. Θα πρέπει να του στείλουμε νέο αλγόριθμο. Απλώ να τον εγκαταστήσουν και η αλλαγή γίνεται εύκολα. Αυτά συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Κατά τα άλλα, πω προκύπτει η φοροδιαφυγή, αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αν του δίνουμε εμεί τι πληροφορίε, Πού είναι ο κίνδυνος, πώς αποφεύγουν το του τις εταιρείε ή τη φοροδιαφυγή. Το θέμα αυτό θα ανακύπτει από καιρού καιρών στο μέλλον. Τι ακούμε όμω από τι εταιρείε. Οι εταιρείε αυτέ που φοροδιαφεύγουν έχουν το πρόβλημα ε, γιατί αν τώρα αποφεύγουν τους φόρους και δεν πληρώνουν το κράτος, αύριο θα πληρώνουν εσά. Ο κίνδυνος λοιπόν είναι παρκτός. Εάν όλοι δουν τον κίνδυνο και τον καταλάβουν, σταματάει και η φοροδιαφυγή. Και τα πράγματα βελτιώνονται για όλους. Και για την τελευταία ερώτηση, Ισχύει μάλλον περισσότερο για την αστυνομία από ότι για την εφορία. Αλλά δεν ξέρω ποιο είναι ο μέσο όρο που δείχνει ότι πληρώνουν περισσότερου φόρου από εμά. Αλλά ελπίζω ότι σήμερα δεν χρειάζονται αυτού του είδου τα μεγάλα δεδομένα, τη πληροφορία για να υπολογίσουν του φόρου ή για την ανάλυση κινδύνου. γιατί αν προσέξετε αυτό που σας έδειξα, είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσει κανείς ότι όλα πάνε καλά, αλλά μπορεί το να έχει κανείς σαν ένα κακοκοινομάλης να κίνδυνος. Πώς επιλύεται αυτό. Κουρεύεται. Είναι τόσο ανόητη η ιδέα. Ευχαριστώ. Κύριε Σάβημα. Σας ευχαριστώ. Και εγώ θα απαντήσω στις ερωτήσεις περίπου στη σειρά με την οποία υπευλήθησαν. Ναι, μοιραζόμαστε ε, τα δεδομένα και με άλλες υπηρεσίες επιβολή του νόμου. Μερικές φορές μέσω των ε, συστημάτων ε, πληροφορικής Ε, όπως είπε και ο, ο συνάδελφός μου, εμείς έχουμε δικαιώματα βάσει των δικαιωμάτων πρόσβασης ε, που έχει κάθε υπηρεσία. Έχουμε καλή συνεργασία με το Πολυτεχνείο του Ταλίν που μας βοηθάει υποβάλλοντας κάποιες λύσεις όσον αφορά τα big data ε, αλλά δεν έχουν, ε, δεν έχουν ε, πρόσβαση στα, στους φακέλους. Έχουν μόνο τη δυνατότητα να μας δώσουν κάποιες πληροφορίες. Επίσης, η ανταλλαγή δεδομένων μερικές φορές εξαρτάται από τα αιτήματα που λαμβάνουμε. Όλες οι ανταλλαγές πάντως, πώς να σας το πω, γίνονται βάσει του τι ζητάει ο καθένας, ποιος είναι ο σκοπός του αιτήματο κλπ. Παρ' όλα αυτά, Υπάρχει και μία ειδική επιτροπή στο κοινοβούλιο μας που ασχολείται με θέματα επιτήρησης και ανείχνευσης στοιχείων. Επιτήρηση και όσον αφορά τις ε, αρχές ασφαλείας όσον αφορά και τις δραστηριότητες της πληροφορίας συμπεριλαμβανομένων και των συλλεγισών πληροφοριών. Εξαρτάται, εξαρτάται. Εμείς έχουμε σαν αστυνομία πολλών ειδών αποθηκευμένες ε, πληροφορίες. Όσον αφορά τώρα τα στοιχεία τα οποία συλλέγονται από διάφορες ε, πηγές, η κύρια ε, δυσκολία είναι η τεχνικής φύσεως, δηλαδή πώς μπορούν να ταξινομηθούν καλά και πώς μπορούν να ενταχθούν σωστά όλα αυτά τα στοιχεία που είναι κατακαιρματισμένα. Ε, μπορεί να έχουν ενδεχομένως κάποια ε, κοινά στοιχεία ή κοινέ διατυπώσεις, αλλά το περιεχόμενο να είναι εντελώς διαφορετικό. Η εργασία λοιπόν η οποία απαιτείται ε, είναι μακρά και δύσκολη. Και ίσως αυτό αποτελεί και μια απειλή σε σχέση με το κατά πόσον είναι σωστά τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται για την λήψη απόφασης, πόσο συχνά γίνονται οι έλεγχοι των στοιχείων αυτών. Ενδεχομένως αυτό που γίνεται στην Εστονία να μην μπορεί να γίνει σε μεγαλύτερες χώρες Ίσως αυτό το σύστημα να είναι πιο εύκολο για μας που είμαστε μικρή χώρα ε, και έχουμε ε, μικρή αστυνομική δύναμη, περίπου 4.000 είναι τα άτομα. Ίσως λοιπόν το μοντέλο να μην είναι σωστό για μεγαλύτερες χώρες και πολυμελέστερες αστυνομικές δυνάμεις πρέπει να σας πω ότι εμείς παρακολουθούμε και τα μέσα κοινωνικής ε, δικτύωσης. Ε, έχουμε αστυνομικούς, ε, αξιωματικούς αστυνομίας που παρακολουθούν τις δραστηριότητες αυτές έτσι ώστε να διαπιστώσουν αν υπάρχουν δραστηριότητες οι οποίες είναι παράνομες ας πούμε κατά νέων ή παιδιών. και επομένως να αναλαμβάνεται δράση έτσι ώστε να προστατευτούν τα δικαιώματα των ε, ανηλίκων. Το ερώτημα που θέσατε είναι κατά πόσον ε, ε, αυτού του είδους οι κανόνες μπορεί να οδηγήσουν σε επικινδυνότητα. Κοιτάξτε, εμείς λέμε ότι ότι όλα τα στοιχεία τα οποία παίρνει η αστυνομία είναι ελεγμένα στοιχεία. Και εάν έχουμε κάποια στοιχεία τα οποία δεν είναι απόλυτα ε, ελεγμένα, τότε θα κάνουμε έναν έλεγχο όλων των connections ε, έτσι ώστε να δούμε κατά πόσον ε, τα στοιχεία είναι σωστά. Μερικές φορές μπορεί να μην λειτουργήσει το σύστημα, αλλά πάντως το θέμα των ιδιωτών δεν είναι μεγάλο πρόβλημα. Εμείς δουλεύουμε και με το Πανεπιστήμιο του Τάρτου Και όντως πρέπει να υπάρχει ένας βαθμός εμπιστοσύνης. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε όλα τα στοιχεία, αλλά τα εμπιστευόμαστε. Ε, ο καθένας από τον οποίο παίρνουμε στοιχεία ε, ε, παίζει και ανάλογα με το βάρος της αξιοπιστίας που έχει. Αλλά σας ξαναλέω, η Εστονία είναι μικρή. και τα στοιχεία τα οποία ε, χρησιμοποιούμε βεβαίως ε, έχουν ένα μικρό περιθώριο στατιστικού σφάλματος, αλλά σε γενικές γραμμές είναι σωστά. Και είχα και μια τελευταία ερώτηση για τους αλγορίθμους, για τα big data και τις ε, δυνατότητες που σχετίζονται. Νομίζω ότι οι αλγόριθμοι των big data έχουν ίδιο βαθμό αξιοπιστίας περίπου με οποιοδήποτε άλλο ερευνητικό εργαλείο. Υπάρχουν καλοί ερευνητές και υπάρχουν και ερευνητές που δεν είναι και πολύ καλοί. Υπάρχουν έρευνες και ερευνητές που βασίζονται σε καλά στοιχεία και σε επιστημονική επαγγελματική προσέγγιση και άλλες όχι. Το πρόβλημα είναι λοιπόν ε, παρόμοιο. Τώρα, το εάν είναι αλγόριθμος ή εάν είναι έρευνα, ε, στην ε, διερεύνηση αδικημάτων εμείς ε, λαμβάνουμε υπόψη όλα τα στοιχεία. Νομίζω λοιπόν ότι η προγνωστική αστυνομική εργασία είναι σημαντική όσον αφορά ορισμένες συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων, αλλά δεν μπορεί καλά να χρησιμοποιηθεί για τα άτομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Η πρώτη απάντηση για τους ε, ιδιωτικούς πολιτές, η είναι μια η υπηρεσία η, οποία η που χρησιμοποιείται σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο. Ε, χρησιμοποιήθηκαν πέρσι δημόσια δεδομένα για να υπολογιστεί κατά πόσον οι μετανάστες ήταν επικίνδυνοι και ε, είχαν κίνδυνο να είναι τρομοκράτες. Το δεύτερο στοιχείο αφορά τον κίνδυνο, αυτό που ανέφερε ο Γιάνν Αλμπριχτ. Περιπτώσεις όπου, για παράδειγμα, το χρώμα των μαλλιών σου θα μπορούσε να προβλέψει την εγκληματική σου ε, διάθεση. Το παράδειγμα που σας ανέφερα για την πρόβλεψη των, των χαρακτηριστικών του. Η πρόγνωση της ε, προσωπικότητας βάσει τα likes στο facebook έχει φανεί την ακριβή σε κάποιο συγκεκριμένο πλαίσιο. Υπάρχουν λοιπόν εκατομμύρια data points και γίνεται ε, αξιολόγηση βάσει του Facebook και των likes του μου. Για παράδειγμα, κάποιος ε, που του αρέσει η Britney Spears μπορεί να είναι πιο πιθανό να είναι ομοφυλόφιλος, νευρωτικός κτλ. Και αυτό μας οδηγεί στο θέμα του κινδύνου. Η προσωπικότητα ακούγεται ε, κάτι πολύ αθώο, αλλά για παράδειγμα το κατά πόσο κάποιο είναι ανευρωτικό. Μπορεί να προβλέψει κατά πόσο έχει ψυχική ασθένεια. Αυτό είναι πάρα πολύ ευαίσθητη πληροφορία και τα Facebook likes μπορεί να θεωρούνται προστατευμένε πληροφορίε και προστατευμένα δεδομένα ακόμα. Υπό την έννοια ότι δεν διατίθενται στου πάντε. Αν κάνει κανεί παρόμοιε προβλέψει και έχουν γίνει τέτοιε προβλέψει από άλλε πηγέ δεδομένων όπω είναι τα δεδομένα κινητών τηλεφώνων γίνουν συσχετισμοί για την φραγκιότητα του ατόμου βάσει του πόσο συχνά απαντά στο τηλέφωνο. Αυτά. Σε τι σημαίνουν ότι ενδεχομένω πάρα πολύ ευαίσθητα δεδομένα είναι προσβάσιμα σε οποιοδήποτε έχει πρόσβαση στα δεδομένα αυτά. Για παράδειγμα, τηλεφωνική εταιρεία, για το Twitter, για παράδειγμα, αν υπολογίζουμε πόσο συχνά τουιτάρει κάποιο και κάνουμε συσχετισμού. Αυτό τι σημαίνει, ότι οποιοδήποτε είναι στο Twitter ουσιαστικά παρέχει αυτά τα ευαίσθητα στοιχεία για τον εαυτό του και παρά το γεγονό ότι υπάρχει μια επιστημονική βάση για τα θέματα αυτά, υπάρχουν και πάρα πολλέ πιθανότητε να είναι ανακριβεί αυτέ οι προβλέψει. Αν οι προβλέψει λοιπόν αυτέ, τι σημαίνει, ότι σε κάποιε βάσει δεδομένων μπορεί να υπάρχουν πολλέ πιθανότητε ε, καθένας μας εδώ στην αίθουσα να είναι σε μια βάση δεδομένων καταχωρισμένος ως νευρωτικός, ως αξιόπιστος και ούτω καθεξής. Και το πρόβλημα είναι ότι είναι δύσκολο να εντοπίσουμε πού βρίσκονται αυτές οι βάσεις δεδομένων, πώς έχουν γίνει οι προβλέψεις και να τις διορθώσουμε σε περίπτωση που είναι ανακριβείς. Αυτό ήταν το ένα στοιχείο που θέλω να αναφέρω. Ένα άλλο θέμα. Δεν έχουμε επιλογή, είπε κάποιος Νομίζω ότι πολλά μπορούν να γίνουν, πολλά μπορούμε να κάνουμε και πολλά παίρνουν από το χέρι μας. Η διαφάνεια δεν είναι ε, λύση για τους λόγους που ανέφερα και προηγουμένω. Και όταν απομακρυνθούμε από τα social media και σκεφτούμε το διαδικτύο των πραγμάτων, υπάρχει εδώ μια στιγμή μεγάλης ευκαιρίας. Έχουμε τις ε, Απειλέ στην ασφάλεια και το privacy και πραγματική ανάγκη να σταματήσει η εκμετάλλευση των δεδομένων. Αυτή είναι η γενιά των δεδομένων που δεν έχουν να κάνουν τίποτα με τους σερβερ. Και μου άρεσε και η κούκλα που χρησιμοποιήθηκε, γιατί είναι σαφές ότι πρόκειται για ένα αντικείμενο το οποίο χρησιμοποιούμε μέσα στα σπίτια μας και δημιουργεί και παράγει στοιχεία. Δεν έχει να κάνει τίποτα αυτό με τους σερβερ που χρησιμοποιούνται ο καταναλωτή δεν ξέρετε τι δεδομένα συλλέγονται, δεν υπάρχει οποιοδήποτε τέτοιο δικαίωμα. Δεν μαθαίνει σχεδόν ποτέ κανεί ε, ότι συλλέγονται τα δεδομένα αυτά για να προβεί σε καταγγελία. Να σταματήσει λοιπόν η εκμετάλλευση των δεδομένων. Αυτό ήταν το πρώτο θέμα. Κατά δεύτερον, υπάρχει ένα έλλειμμα σε ό,τι αφορά την εφαρμογή. Και πάλι το παράδειγμα που ανέφερα από την Cambridge Analytica από τη ΣΥΠΑ. Πώς ε, μια εταιρεία που έχει την κατρική της ΗΠΑ, αλλά αποτελεί ουσιαστικά βρετανική εταιρεία σε έναν βαθμό. Άρα υπάρχουν πολλές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα το παιχνίδι που είδαμε προηγουμένως, που είναι εντελώ και παντελώ παράνομες. Και επειδή υπάρχει πρόβλημα στην εφαρμογή της νομοθεσία και είναι χαμηλό το κόστος για εταιρείας, για να μην συμμορφώνονται στην, με την αυτή. Τέλος, για την Κίνα. Μας απασχολεί πάρα πολύ η Κίνα. Και ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία που είδαμε στις ειδήσει και τρομακτικό μάλιστα, είναι ο υπολογισμό τη φερεγγιότητα των πολιτών, όχι μόνο για να υπολογιστεί η φερικαιότητα του πολίτη, αλλά και το πόσο καλή και ευγενεί είναι ω πολίτε. Αυτό είναι στη φάση σχεδιασμού ακόμα δεν ξέρουμε κατά πόσο στέκει αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι πάρα πολύ ανησυχητικό γιατί είναι παρεμβατικό και επίση είναι πάρα πολλέ οι πιθανότητε να υπάρχει ανακρίβεια στην υπολογισμό αυτό. Και τέλο, για την εφαρμογή του δικαίου, την επιβολή του δικαίου. Γιατί σα έδωσα αυτό το παράδειγμα για την Cambridge αναλυτικά, γιατί περιλαμβάνεται μεγάλο ε, ποσοστό μύθου σε ό,τι αφορά τα big data. Η ακρίβεια που θεωρείται ότι υπάρχει δεδομένου ότι πολλοί πιστεύουν ότι μπορούν να επιλύσουν τα big data προβλήματα που δεν μπορούν να επιλύσουν. Και γι' αυτό λοιπόν ότι θα μπορούσαμε να βασιστούμε στις ε, προβλέψεις αυτές χωρίς ε, περαιτέρω έρευνα. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Και επίσης υπάρχει και μια διαφορά μεταξύ των προβλέψεων που γίνονται βάσει τόπου και βάσει ατόμου. Ακόμα και χρησιμοποιηθούν αστυνομικά στοιχεία, τα αστυνομικά στοιχεία, ο φάκελο στην αστυνομία είναι κάτι το προληπτικό. Παραλαμβάνει και παρουσιάζει ε, τι αναφορέ τη αστυνομία. Ε, κάποια εγκλήματα αναφέρονται ως ίσονος σημασίας, κάποια ως μεγαλύτερη σημασίας και το καθεξή. Και επίση ε, σε ό,τι αφορά την πρόβλεψη και την, ε, την πρόβλεψη των εξελίξεων, αν βασιστούμε αποκλειστικά στα αστυνομικά στοιχεία, μπορεί να καταλήξουμε σε ένα ανακριβές αποτέλεσμα. Σε ό,τι αφορά λοιπόν ε, ε, τι προβλέψει που αφορούν ένα άτομο, δεν θα πρέπει να γίνεται κάτι τέτοιο ακριβώ επειδή είναι τόσο μεγάλο ο κίνδυνο ανακριβία. Okay. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ τους ομιλητές. Ευχαριστώ που ανασκουμπόθηκαν και απάντησαν στις ερωτήσεις. Βλέπω ότι ο κύριος Ρίστερ θέλει το λόγο. Ε, έχει τη δυνατότητα, διότι χρόνος υπάρχει. Σας δίνω λοιπόν το λόγο και μετά πάλι στην Άννα Γκόμες. Για μια παρατήρηση. Ναι, με συγχωρείτε απλώς ε, να μιλήσω για το θέμα της βαθμολόγησης των στατιστικών ε, εντύπων. Είναι πολύ περίπλοκες διαδικασίες και η βαθμολόγηση, όπως είπατε, δεν αντεύουν κατά 100% αν είστε ομοφιλόφιλος ή πάντρελος, ε, δίνουν ένα ποσοστό από 1 έως 100. Ωστότε, με, οπότε μετά το θέμα είναι όταν παίρνει κανείς στα χέρια του αυτό το ποσοστό, το κάνει. Η αστυνομία, εως 100 τότε με οποτε μετα το πάρει, ίσως υπάρχει πιθανότητα να το αξιοποιήσει. Ή υπάρχει πιθανότητα στον εμπορικό κόσμο να θεωρήσει κανείς ότι εγώ θα αγοράσω τσίχλες άμα βγω από αυτό το κτίριο, ας πούμε, θα είναι η πρώτη μου κίνηση. Αυτές οι μέθοδοι χρησιμοποιούνται, αλλά το κτιριο α είναι πώς τις χρησιμοποιεί κανείς. Πώς τις χρησιμοποιούν οι στατιστικολόγοι, μαθηματικοί, οι επιστήμονες, εξαρτάται από την τεχνογνωσία τους και πόσο αυστηρά θεωρήσουν τον αλγόριθμο για να παράξουν τα αποτελέσματα που θέλουν. Οπότε ναι, ίσως τα υψηλά ποσοστά, πιθανότητα ότι μπορεί να αγοράσω κάτι τώρα ας πούμε, μπορεί και να έχει σχέση με το ότι τα πράγματα δεν έγιναν όπως έπρεπε. Δεν συμφωνώ λοιπόν ακριβώς ότι γίνονται λάθη. Προφανώς γίνονται σε ένα βαθμό, όμω η βαθμολόγηση είναι αυτή που έχει σημασία. Δεν είναι δεσμευτική κάποια οριακή αξία. Ευχαριστώ. Ναι. Προφανώς, η κυρία Κάλ Τέινερ προφανώς μπορεί να απαντήσει, αλλά να τονίσω ότι σημαντικό είναι και πώς προγραμματίζει κανείς τους αλγορίθμους. Διότι λόγω χάρη απόφαση για το τι θα θέσω ως ιδιότητα του καλού πολίτη στο βαθμολόγιο των πολιτών στην Κίνα, το αν κάποιος καπνίζει ή όχι, εάν κάποιο την νύχτα την τάδε ώρα βγαίνει από το σπίτι του ή όχι και ούτω καθεξής, είναι πολύ αυθαίρετο. Κυρία Καλτένε, γνωρίζω ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ βαθμολόγησης και κατάρτισης προφίλ. Και επίσης πολύ καλά γνωρίζω ότι κανένας αλγόριθμος, κανένα, κανένα ποσοστό δεν λειτουργεί ω μονόδρομο για το αν είναι κανεί αξιόπιστο ή όχι. Παρ' όλα αυτά, από την οπτική γωνία του καταναλωτού ή πολίτη, η βαθμολόγηση, όπω λέτε, είναι ιδιαίτερα περίπλοκη. Χρησιμοποιεί τεράστιο όγκο δεδομένων. Και τα ζεστήματα βαθμολόγηση επηρεάζει τις αποφάσεις σε σχέση, ο υπολογισμό επηρεάζει τι αποφάσεις σε σχέση με τους ανθρώπους. Εάν κάποιο, ας πούμε μπορεί να προσληφθεί ή όχι, ή αν εργάζεται σε έναν τομέα με χαμηλό εισόδημα. Ας πούμε ότι είμαστε σε μια προκήρυξη για μια θέση με χαμηλή αριμαγή και χιλιάδε υποβάλλουν αίτηση. Εκεί μπορεί να παίξουν ρόλο τα ποσοστά ή το ιατρικό προφίλ των ανθρώπων από τα μεγάλα δεδομένα. Δηλαδή κάποιο ορίζει αξίε που είναι κάπω αφαίρετε για το τι είναι ο καλό υποψήφιο και ο αλγόριθμο, οι μηχανισμοί αυτοί που λειτουργούν σαν ένα από ένα μαύρο κουτί, τελικά δίνουν πολύ συγκεκριμένα αποτελέσματα. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αν υποψήφιο διαρκώ δεν παίρνει τη θέση εργασία την αποβάλλει τα χαρτιά του και δεν ξέρει πώ λειτουργεί το σύστημα, δεν ξέρει ποια είναι αυτά τα σημεία στο σύστημα που ε, επιτρέπουν να γίνεται η διαλογή, αν είναι ακριβή ή όχι, αυτό είναι ακριβώ το πρόβλημα. Δεν είναι η ακρίβεια των αλγορίθμων ή η καλύτερη ποιότητα των δεδομένων. Αυτό είναι ένα θεμελιώδε πρόβλημα. Υπάρχει έλλειψη ισορροπία εξουσία μεταξύ των κέντρων που λαμβάνουν τι αποφάσει και των ανθρώπων που θέλουν απλώ να ζήσουν τη ζωή του. <coughs> Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι αυτό δείχνει ότι ακριβώ πρέπει να το μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα στο μέλλον και αυτό που κάνουμε εδώ είναι να προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε τη διαδικασία. Ε, έχουν ήδη γίνει πολλά και η Άννα Γκόμες έχει αναλάβει την ε, ε, πρωτοκαθεδρία στο να μας οδηγήσει στη σωστή κατεύθυνση. Σε παρακαλώ, Άννα, να σου δώσω το λόγο για σύντομες καταληπτές παρατηρήσεις. Δεν είμαι στην πρωτοκαθεδρία. Στην πρώτη θέση των μαθητών είμαι. Στο πρώτο θρανείο. Όπως είπες, αυτό είναι μια πορεία στο χρόνο. Συζητώντας με τους ενδιαφερόμενους και τους φορείς, βλέπουμε μεγάλους κινδύνους πέρα από τα μεγάλα ωφέλη. Και αυτούς τους μεγάλους κινδύνους βλέπουμε, τους βλέπουμε να αυξάνονται και θα πρέπει να τους μειώσουμε όσο μπορούμε. Από όσα άκουσα, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούμε να βασιστούμε σε κανένα σύστημα με επιμέρους κατακαιρματισμένες αποφάσεις ή ε, με ε, διαδικασία λήψης αποφάσεων όπου να υπάρχει και λογοδοσία. Οι αποφάσεις λαμβάνονται από διαφορετικούς ηθήνοντες σε διαφορετικά επίπεδα με οποιαδήποτε ιδιότητα μπορεί να φανταστεί κανείς. Ιδάλλως, οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές. Όχι μόνο για τις δουλειές λόγου χάρη που μιλάγαμε πριν, με βάση το παράδειγμα που δόθηκε, αλλά στον τομέα των σπιτιών των κατοικιών, στο στεγαστικό δηλαδή, στα ποινικά, στα... σε ό,τι αφορά τα δικήματα, το δίκαιο. Η άλλη πτυχή είναι ότι το ζωτικό ερώτημα για τις ε, αρχές της διοκτικές είναι ότι να έχουμε τους καλύτερους επαγγελματίες και να επενδύσουμε στο να έχουμε τους καλύτερους επαγγελματίες και στα καλύτερα όμως πρότυπα μαζί για να αντιμετωπίσουμε την ενδεχόμενη κακοχρησία ή την, ε, τις, τις αυλεψίες μάλλον σε ε, εγκληματικές απόπειρες ή ενέργειες. Είναι πάρα πολλά αυτά που θα μπορούσα να αναπτύξω, αλλά τώρα δεν είναι ανάγκη να τα συνοψίσω έτσι, βιαστικά. Σίγουρα ήταν πολύ χρήσιμη η συζήτηση και πραγματικά αναμένω διακαώς τις συνεισφορές σας αυτές που εσείς και όλοι οι υπόλοιποι θα μπορούσατε να μας αποστείλετε. Όπως είπε και ο Άλμπερτ, αυτό είναι η αρχή μιας διαδικασίας, η αρχή ενός ταξιδιού. Όπου αρχίζουμε επιπλέον να αντιλαμβανόμαστε τις επιπλοκές όλου αυτού του φαινομένου. Εμείς ως Επιτροπή δεν θέλουμε να μείνουμε πίσω. Να μείνουμε πίσω στην όλη μάχη για την προστασία των θεμελιωδών δικαιωμάτων. Αυτό είναι το βασικό στοιχείο. Ένα στοιχείο που ήδη καλύπτει ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία των Δεδομένων ε, και εκεί που χρειάζεται να εντοπίσουμε τα προβλήματα, τα κενά, τις ελλείψεις, τους ε, συμπληρωματικούς κανόνες, ίσως όχι κανονισμούς αυτή τη στιγμή, αναγκαστικά, αλλά τις αλλαγές της συμπεριφορά στην κουλτούρα που ίσως ε, επιβάλλονται. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και πάλι όλους μας τους ομιλητές και βεβαίω και όλου του υπόλοιπου, όσου συνεισέφεραν σε αυτή την εκδήλωση. Σας εύχομαι μια πολύ όμορφη βραδιά. Θα το ξαναδούμε πολύ σύντομα το θέμα. Ευχαριστώ.